Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μα με την παραδοσιακή καθυστέρηση τη Δευτέρα, που είναι μια δύσκολη μέρα για να έλθουν εγκαίρω οι συνάδελφοι στη συνεδρίαση. Αν δεν έχετε παρατηρήσει ε, για την ημερήσια διάταξη, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Υποδεχόμαστε σήμερα δύο προσκεκλημένους, ε, τον ε, αντιστράτηγο Βαν Ως, Γενικό Διευθυντή του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις 4.30 θα έχουμε μαζί μας ε, τον κύριο Σιμούνοβιτς, Υφυπουργό, στο Υπουργείο Μήνας της Δημοκρατίας της Κροατίας. Σας υπενθυμίζω ότι εκτάκτος τη Δευτέρα κατά την συνεδρίαση της Ολομέλειας του Στρασβούργου θα διοργανώσουμε μια έκτακτη ε, συνεδρίαση στις 7 τη Δευτέρα γιατί θα έρθει ο στρατηγός Αμπριάλ για την μεταρρύθμιση του ΝΑΤΟ στο Νόρφολκ, είναι ο επικεφαλής. Θα έρθει λοιπόν και έτσι μετά την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί τους στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Στρασβούργου. Θα δώσω αμέσως λοιπόν το λόγο τώρα στον στράτηγο Βαν Ως που αντικατέστησε τον στρατηγό Λίκη που πολλές φορές ε, είχε έρθει στην υποεπιτροπή μας και είχε μιλήσει. Θα είναι επικεφαλής λοιπόν, ε, μάλλον είναι επικεφαλής από τις 28 Μαΐου 2010 του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Υπάρχουν ζητήματα που άπτονται του πεδίου αρμοδιοτήτων σας και θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε σήμερα. Ένα από αυτά βέβαια είναι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η τελευταία χρονολογικά, την οποία δεν έχουμε συζητήσει ακόμα ε, για τη Σομαλία, ε, στην Ουγκάντα συγκεκριμένα αναπτύσσεται αυτή η επιχείρηση, τις δυνατότητες, ένα, πρόγραμμα, ένα πρόβλημα που επανέρχεται επανειλημμένος, θα θέλαμε να δούμε και τους στόχους τους γενικούς 2010. Επίσης η υλοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας, η εφαρμογή της, το συζητούμε πολλές φορές και στην Επιτροπή Εξωτερικών και στην Επιτροπή μας εν μέρη για την ΕΕΔ, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και θα ήθελα να μας πείτε και εσείς πού εντάσσονται στην αρχιτεκτονική της υπηρεσία αυτής οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και βέβαια η σφαιρική προσέγγιση, η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία, ένα θέμα πολύ αγαπητό σε εσά όπως γνωρίζω και το οποίο το έχουμε συζητήσει και εμείς πολλές φορές στην Υποεπιτροπή μας και δει με την έκθεση του Κριστιαν Λέρ, του συναδέλφου μας. Στρατηγέ μου, σας δίνω το λόγο. Thank you very much for this kind introduction. Uh, σας ευχαριστώ για την ε, θερμή αυτή υποδοχή. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα και να μιλώ με τα μέλη σας, το οποίο μου δίνει και την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε και τις δικές μας ιδέες. Και φυσικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μας να ακούσω, για μένα να ακούσω τις δικές σας ιδέες για να καταλήξουμε στους καλύτερους τρόπους ε, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας. Όπως εξήγησε και ο Πρόεδρος, Είμαι διάδοχος ε, του στρατηγού Λίκη ως Γενικός Διευθυντής ε, του Στοχητικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω δύο λόγια για το ρόλο μου, γιατί έχετε συναντηθεί με τον στρατηγό Σιρενίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής. Εγώ είμαι Γενικός Διευθυντής του Στρατιωτικού Επιτελείου. Ποια είναι η διαφορά. Εγώ είμαι επικεφαλής του στρατιωτικού επιτελείου εντός των ευρωπαϊκών δομών με καθήκον να, υποστηρίξω, να υποστηρίζω την Στρατιωτική Επιτροπή. Συχνά μου μιλάνε λες και είμαι ο υπουργό Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν αληθεύει. Ε, είμαι στην υπηρεσία των 27 κρατών μελών και αυτοί απαρτίζουν ε, όπως και ο στρατηγός Σιρέν, το, Στρατιωτική Επιτροπή. Δύο. Διτός μάλλον είναι ο ρόλο μου. Υποστηρίζω την Στρατιωτική Επιτροπή και την... Ε, παρέχουμε σε πολιτικό επίπεδο στρατιωτικές συμβουλές. Αν υπάρξει απόφαση να χρησιμοποιηθεί ο στρατός, στην περίπτωση αυτή, εντός των ε, δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενταχθούμε από 1η Ιανουαρίου στην Υπηρεσία εξωτερική δράση. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, καθήκον μου είναι να διασφαλίσω την εφαρμογή του σκέλους αυτού σε συνεργασία με το πολιτικό σκέλος, με τις υπόλοιπες δομές. Και ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να καταλάβω τη θέση αυτή και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που την κατέχω από τον Μάιο του τρέχοντος έτους είναι γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ε, συναρπαστικό για ένα στρατιωτικό στον καιρό μας να ανήκει στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω υπηρετήσει στο ΝΑΤΟ και στο ιστορικό του ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα ο στρατός ζητάει και από άλλα σκέλη να διαδραματίσουν το ρόλο τους στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Εμείς κατανοούμε ότι το στρατιωτικό σκέλος δεν μπορεί από μόνο του να επιλύσει κρίσεις. Πάντα θα πρέπει σε στενή συνεργασία να ακολουθούμε μια συνολική προσέγγιση μαζί με όλους τους υπόλοιπους φορείς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι έχουν γίνει πολύ σοφά βήματα προς μια τέτοια συνολική ε, προσέγγιση, το ονομάζουμε ΚΕΠΑ, ξέρετε τι περιέχει αυτό, και μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας ε, δημιουργούμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και αυτό σας είναι γνωστό. Το πιο θετικό στοιχείο θεωρώ σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι ότι θα αυξήσει τις δυνατότητες για μια συνολική προσέγγιση μια δομή ακόμα πια ευρεία από την ΚΕΠΑ. Ο κ. Κλοπανάουρη είναι φυσικά πολύ καλός μου συνάδελφος. Και με την επικεφαλής του CNPD συνεργαζόμαστε στενά. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε μια μεγάλη βελτίωση γιατί ξέρετε την τελευταία δεκαετία ασχολούμαι με στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα θα έχουμε την υπηρεσία εξωτερική δράση η οποία θα καταστήσει δυνατόν να υπάρξει ακόμα και μια πιο ευρεία προσέγγιση. Γιατί, αυτό ελπίζω τουλάχιστον, θα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε σε στενότερη συνεργασία και με τα όσα πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σέβομαι ιδιαίτερα την Επιτροπή και έχουν σημαντικά μέσα τα οποία και αξιοποιούν σε πολύ σημαντικούς και δύσκολους τομείς για την αντιμετώπιση των κρίσεων, για την απτυξιακή βοήθεια και το καθεξής. Ξέρετε και εσείς πολλά από τα προγράμματα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ε, συνεργαστούμε και να καταβάλουμε από κοινού προσπάθειες. Δεν σημαίνει αυτό φυσικά ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα συντονίζει τα πάντα, θα διατηρήσει το ρόλο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω. ότι υπάρχει κάποιο λόγο που ονομάζεται η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο ε, Υπουργό Εξωτερικών, κοιτώντα τα καθήκοντά τη και κοιτώντα και τι γίνεται στα κράτη-μέλη, φυσικά θα διαθέτει τα δικά τη μέσα και συμπεριλαμβάνονται και οι υποδομές της ΚΕΠΑ, αλλά πέραν από αυτό θα συντονίζει και τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες. Ξέρετε τι έχουν αποφασιστεί, τι έχει αποφασιστεί για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Πέραν αυτών όμως θα χρησιμοποιεί και την τεχνογνωσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική βελτίωση οι συντονιστικοί μηχανισμοί, όπως θα έκανε και ένας υπουργό εξωτερικών παρεπιπτόντος και σε μια κυβέρνηση. Δεν είναι αφεντικό των υπόλοιπων υπουργών. Έτσι και η υπατή εκπρόσωπος θα έχει τη δική της υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αλλά μπορεί να λαμβάνει και πρωτοβουλίες συντονισμού με άλλους φορείς. Και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι υπάρχουν αυτοί οι φορείς, οι οποίοι μπορούν να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντική σε πολλούς τομείς, αλλά και στον τομέα της άμυνας και της ε, ασφάλειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θεωρώ. Και θα ήθελα να σημειώσω μία ανησυχία μου. Ξέρω ότι πολλά μέλη της Επιτροπής αυτής ή πολλά κράτη-μέλη ανησυχούν και λένε ότι μέσα σε αυτήν την ευρεία δομή το στρατιωτικό σκέλος θα είναι τόσο περιορισμένο που μπορεί να μην έχει σημαντικό ρόλο. Να σας πω ότι εμένα αυτό δεν με ανησυχεί. Πάντα ζητούσαμε μια τέτοια συνολική προσέγγιση και με τον Άτο. Και το συζητάμε αυτό μάλιστα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό επιτέλους γίνεται και προβλέπω ότι και το στρατιωτικό σκέλος θα αναδειχθεί πιο επιτυχές χάρη σε αυτή την συνολική προσέγγιση. Μαζί με όλα τα άλλα, τα πολιτικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχουν τεθεί και κάποια ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη θέση της υπηρεσίας εσωτερικής δράσης και τη θέση του και σκέλους στο εσωτερικό της δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία. Το έχουμε συμφωνήσει ιδιαίτερα ήδη με, τον, την υπατή εκπρόσωπο. Και όλοι, και το Συμβούλιο και ο στρατηγός είναι ξεκάθαρος. Αν υπάρξει κρίση, η ύπατη εκπρόσωπος θα καλέσει σε στρογγυλή τράπεζα τους ε, αρμόδιους φορείς που είναι αρκετοί, αλλά σίγουρα σε αυτούς τους φορείς θα συγκαταλέγεται και το, ο στρατός. Και θα Παρέχουμε λοιπόν τις συμβουλές μας, αν ούτως αποφασιστεί. Αν πρόκειται για μια απόφαση που προαπαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο, θα συμμετέχουμε κι εμείς στην διαδικασία λήψης της απόφασης. γιατί όταν χρησιμοποιείται ο στρατός πρέπει, θεωρώ, να δώσει τη γνώμη του και ο ίδιος ο στρατός, κατά πόσον είναι εφικτά τα σχέδια και όχι ευσεβείς πόθη. Και άλλος ένας λόγος που χρειάζεται η εμπλοκή του στρατού είναι ότι αντικαταπλίζεται πάντα η εθνική κατάσταση. Ξέρω ότι είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση και την έχετε ήδη κάνει και στο παρελθόν, αλλά θα την κάνετε και στο μέλλον επανειλημμένα σε ό,τι αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα έχω υποχρέωση αναφοράς και στα Εθνικά Κοινοβούλια, αν μου το ζητήσει κάποιο Εθνικό Κοινοβούλιο, για την στρατιωτική συνδρομή του εκάστοτε κράτους. Είμαι υπόλογο αυτούς και φυσικά είμαι υπόλογο και θα χαρώ να απαντήσω και στις ερωτήσεις ε, της τη Επιτροπή Υποσχέθηκα ότι θα μιλήσω μόνο 15 λεπτά. Να πω δύο λόγια για τις τρέχουσες ε, επιχειρήσεις και για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας, ίσως και δύο λόγια και για τον ΝΑΤΟ. Για τις τρέχουσες ε, επιχειρήσεις. Όλοι γνωρίζετε, νομίζω, τις πιο σημαντικές πτυχές. Αλθεία. Επιχείρηση Αλθεία στην ε, Βοσνία Ζεργοβίνη. Δύο χρόνια τώρα περίπου αναφέρεται ότι η κατάσταση είναι σταθερή. Ξέρουμε λοιπόν τι έγινε τώρα και με τις εκλογές σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Αποφασίστηκε να, να συνεχίσουμε την εκτελεστική αποστολή. Ήταν πολιτική η απόφαση αυτή που λήφθη. δεν έχουμε αρκετά μέλη για την εκτελεστική αυτή αποστολή, αλλά βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη και σταθερή. Και ο στρατός λοιπόν αποφάσισε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκτελεστική αποστολή, παρά το γεγονός ότι αν φυσικά κάτι ανακύψει, ο κίνδυνος θα είναι μεγαλύτερος, επειδή έχουμε λιγότερα άτομα. Αυτό που είναι σημαντικό, και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γι' αυτό, είναι ότι από 1η Ιουλίου γρηγορότερα δηλαδή από ό,τι προγραμματιζόταν, ξεκινήσαμε μια επιχείρηση εκπαίδευσης για την υποστήριξη των βοσνιακών αρχών. Δεν είναι εκτελεστική αποστολή αυτή. Και μετά από δικό τους αίτημα προβαίνουμε σε εκπαίδευση, κατάρτιση. Οι βοσνιακές αρχές λοιπόν το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να μας ζητήσουν τι θέλουν. Η επιχείρηση Αταλάντα χαίρομαι που μπορώ να σας αναφέρω ότι είναι πολύ επιτυχής η επιχείρηση αυτή. Κοιτώντας τα αριθμητικά στοιχεία, πέρσι είχαμε ...21 επιτυχής ε, παρεμβάσεις. 123 είναι το φετινό νούμερο, 57 εξ αυτών από τη UNAFOR. αλλήλου, συνειδητοποιούμε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, είναι σαφές ότι δεν αποτρέπουμε α, επαρκώς την πειρατεία, γιατί εξακολουθεί να υφίσταται η πειρατεία. Άρα όλο και πιο πολλοί συμφωνούν ότι θα πρέπει να γίνουν πιο πολλά για την ανάπτυξη του δυναμικού μας. Δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσεις, αλλά εγώ υποστηρίζω την γενικότερη σκέψη εντός ε, των δυνατοτήτων μας τα σκάφη της επιχείρησης ήδη το πράττουν αυτό. Εκπαιδεύουν, για παράδειγμα, τις ε, τοπικές αρχές. Αν θέλουμε όμως να έχουμε μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πιο έντονα σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας κατά της πειρατείας και αυτό ίσως να μην είναι το ευκταίο η Ευρωπαϊκή Αποστολή στην Ουγγάντα για την ε, εκπαιδευτική αποστολή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουγγάντα, για τη Σομαλία. Έχει στεφθεί με επιτυχία η εκπαιδευτική αποστολή αυτή. Έχει ολοκληρωθεί πλέον η πρώτη παρτίδα, οι οποίοι ασχολούνται με εκπαίδευση ενσωμάτωσης πλέον και μετά θα αποσταλεί η αποσταλή αυτή στο στο Μογκαντήσου με την υποστήριξη των ΙΠΑ, παραπληκτόντως για να συνδράμουν στο TFG της Σομαλίας και να ενταχθούν έτσι με αυτούς που εκπαιδεύσαμε στην Ουγκάντα. Αυτό δεν είναι... Είναι μάλλον συμφωνία που είχαμε και με την Αφρικανική Ένωση. Για το, πολιτικό, για το στρατιωτικό σκέλος όμως ε, καθήκον μου είναι να εκπαιδεύσω τους εκπαιδευόμενους. Αλλά φυσικά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το κατά πόσο θα ενσωματωθούν σωστά στο TFG οι εκπαιδευόμενοι αυτοί. Γιατί αν ενσωματωθούν σωστά, σημαίνει αυτό ότι ήταν καλή και η εκπαίδευση τους. Και πολλά έχουμε κάνει για να στεφτεί με επιτυχία η ενσωμάτωση αυτή, υπό πολύ δύσκολε συνθήκες μάλιστα. Και σχεδόν έχει περάσει το τέταρτο που έχω στην διάθεσή μου. Να συνεχίσω. Ευχαριστώ. Ανάπτυξη δυναμικού. Um, it's clear. Είναι σαφές ότι φέτος, ιδίως δε του χρόνου, Η βασική εστίαση είναι η επικεφαλής ε, των επιτελείων και η Υπουργή Άμυνας, γιατί με εξαίρεση τρεις χώρες, ε, σε όλες τις περιπτώσεις της υπόλοιπης υπάρχουν τεράστιες περικοπές στον προπολογισμό. Και αυτό βέβαια δεν είναι καλή είδηση. Αυτό όμως όπως γνωρίζετε δεν ισχύει μόνο για το στρατό. Βλέπω ένα θετικό πάντως, ε, ότι δηλαδή υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να δώσουν με μεγαλύτερη προτεραιότητα στη συνεργασία με τα άλλα κράτη-μέλη. Εάν έχεις κάποιες φιλοδοξίες δεν θέλεις να τις μειώσεις, δεν θες να τις ελαττώσεις. Αν λοιπόν θέλεις να έχεις τις δυνατότητες ώστε να φέρεις επέρα στις αποστολές σου, χρειάζεσαι συνεργασία για να μείνεις σε αυτό το επίπεδο δυνατοτήτων. Και μία από αυτές τις δυνατότητε ε, και ένα πολύ καλό παράδειγμα η συνεργασία είναι η γαλλοβρετανική συνεργασία. Άκουσα κάποιες ανησυχίες αν είναι ευρωπαϊκό το σώμα αυτό ή όχι τελικά, αλλά και στην υπουργική, μάλλον στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνα ε, στην Γάνδη, ε, το συζητήσαμε και είπαμε ότι μία από τις δυνατότητες για να συνεχίσουν να υπάρχουν δυνατότητες που δεν μπορεί κάποια χώρα να τις έχει μόνη της, Μία από τις δυνατότητες λοιπόν είναι η συνεργασία. Βέβαια, σε ό,τι αφορά την ε, γαλλοβρετανική συνεργασία υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, μία από αυτές όμως είναι και αυτή και στη συνεργασία ε, υπάρχουν και άλλες προσπάθειες ε, διμερείς, πολυμερείς ε, μεταξύ πολλών κρατών και όταν δημιουργούνται δυνατότητες και υπάρχει βελτίωση, εμένα με ικανοποιεί αυτό. Αυτές οι δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλα διεθνή πλαίσια. Όχι δηλαδή κατά ανάγκη πάντοτε και μόνο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η καλή είδηση όμως νομίζω είναι ότι τουλάχιστον δημιουργούνται ευρωπαϊκές δυνατότητες. Και αν έχουμε ευρωπαϊκές δυνατότητες, αυτό εν μέρει θα καθορίσει και την επιρροή που μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις δυνατότητες ε, που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιλύει κρίση σε περίπτωση που θέλει το πράξει από μόνη της ή σε συντονισμό με άλλους. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα δεν έχουμε όμως ακόμη καταλήξει αποφάσεις. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στον τομέα της ανάπτυξης δυνατοτήτων λόγω ιδίω των περικοπών στον προϋπολογισμό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να απαντήσουμε και ένα άλλο ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πού δίνει προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, τι μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορούν να προσφέρουν ή δεν προσφέρουν άλλοι. Συμμερίζομαι όσους λένε ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε επικάλυψη. Δηλαδή όταν κάποιος θα καταφέρει καλά κάποιοι, γιατί θα το κάνουμε κι εμείς. Κάποιες φορές όμως υπάρχει λόγος βέβαια. Σίγουρα η επικάλυψη βέβαια κοστίζει, ό,τι και να κάνουμε. Τι μπορεί να προσφέρει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιπροσθέτω, επιπλέον. Η απάντηση που έχω να δώσω σε αυτό το ερώτημα ουσιαστικά σχετίζεται με την εισαγωγή που έκανα. Συνολική προσέγγιση. Ένοπλε δυνάμεις σε συνδυασμό με όλους τους άλλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν επειδή ακριβώ υπάρχουν όλα αυτά τα διαφορετικά μέσα μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία μόνο και μόνο οργανώντας αυτή την συνολική προσέγγιση. Ήδη βελτιωθήκαμε πολύ την τελευταία δεκαετία, αλλά σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Σε ό,τι αφορά και το σχεδιασμό και τις διαδικασίες. Μπορούμε επίσης ε, να καταλήξουμε σε περισσότερη συνέργεια και αποτελεσματικότητα. Υπήρξε και μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Δεν το λέω απλά για να είμαι καλός, αλλά με βοήθησε και εμένα στο πώς να περάσω τα μηνύματά μου και στο πώς μπορούμε αυτές τις στρατηγικές ε, να τις ε, περαιτέρω, να τις αναπτύξουμε. Ένα απλό παράδειγμα που μπορώ να δώσω, αν και μπορώ να δώσω και άλλα 20 παραδείγματα πάρα πολύ εύκολα, αν είμαστε στην ίδια περιοχή με στρατιωτικά και πολιτικά μέσα, η πολιτική το πολιτικό σκέλος χρειάζεται ιατρική υποστήριξη. Γιατί να μην έχουμε μια κοινή ιατρική υποστήριξη και με το στρατιωτικό σκέλος. Γιατί, για, μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί να μην έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλήξουμε σε συνέργειες αλλά και σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Λιγότερο κόστος αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο, είναι ένας τομέας όπου πραγματικά μπορεί να υπάρξει προστιθέμενη αξία. Ε, ε, Φυσικά μπορούμε να διευκολύνουμε ε, την κατάληξη ή την, ε, το σχεδιασμό ε, πολιετών, πολυκρατικών σχεδίων. Εμείς φυσικά και πρέπει πρώτα απ' όλα να καθορίσουμε τις δικές μας απαιτήσει, αλλά κάνοντας αυτό μπορούμε να δούμε πρώτον πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και μετά ε, δίνουμε τα σχετικά στοιχεία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, στο EDA, και στη συνέχεια βλέπει αυτός πώς μπορεί να κάνει κάποιους ε, συνδυασμούς, να συνδυάσει την έρευνα, την τεχνολογία των διαφόρων κρατών μελών και με αυτό το συνδυασμό να βοηθήσει την αμυντική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να έχει περισσότερες αγορές. Και νομίζω ότι αυτός μπορεί να είναι ένας πολύ καλός στόχος ίσως και αυτός σκοπός. Τελικά, είναι σαφές ότι εάν είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θα έχουμε και περισσότερες δυνατότητες ε, έχοντας τον ίδιο προϋπολογισμό. Και αυτό είναι σημαντικό. Να μιλήσω για τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγες παρατηρήσεις ε, έχω να κάνω. Είναι ιδιαίτερος χρήσιμο το ότι η Βαρόνια και ο Γενικός Γραμματέας Ράμσμουσεν διακήρυξαν την πολιτική τους φιλοδοξία πολύ ξεκάθαρα για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ μπορώ να πω ότι αυτό σίγουρα δεν είναι κακό. Να υπάρχει δηλαδή αυτή η πολιτική φιλοδοξία και έτσι συνεργαζόμαστε, να συνεργαζόμαστε μάλλον, ώστε να το πιο στενά με το ΝΑΤΟ εκεί που μπορούμε. Βέβαια, δεν είναι τόσο καλό αυτό όσο νομίζουν ορισμένοι, γιατί το πολιτικό πλαίσιο εξακολουθεί να καθορίζεται. ξέρω ότι παραδείγματο χάρη δεν μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Και κάποιε φορέ η συνεργασία καθίσταται δυσχερή. Όλοι βέβαια καταλαβαίνουν ότι από τη στιγμή που 21 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη του ΝΑΤΟ υπάρχουν δυνατότητες να εξασφαλιστεί ότι σε επίπεδο τακτικής και επιχειρήσεων μπορούμε να έχουμε μία δέσμη δογμάτων, διαδικοσιών, ορολογίας κτλ. Διότι αν αυτά διέφεραν αυτό θα είχε καταστροφικές συνέπειες όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν είναι όμως πάντα ο, τρόπο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος συνεργασίας. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει πολιτική φιλοδοξία να βελτιωθεί και αυτό το επίπεδο. Και αυτά νομίζω με αυτά μπορώ να σταματήσω κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ στρατηγέ μου. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους που επιθυμούν να μιλήσουν, αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να επανέλθω σε δύο σημεία, τα οποία έχουν να κάνουν τις επιχειρήσεις και πολύ ειλικρινεί ήσασταν όταν μιλήσατε για την Αταλάντα. Σίγουρα όλοι ε, χαιρετίζουμε την επιτυχία τη επιχείρηση αυτή, ωστόσο ε, συγχρόνως υπάρχουν κάποια αντιφατικά στατιστικά στοιχεία που σημειώνουν αύξηση πειρατικών επιθέσεων. Ε, βέβαια, πολλέ από αυτέ τι αντιμετωπίζουν οι ναυτικέ δυνάμει με επιτυχία. Και υπογραμμίσατε και μπορούμε να μιλήσουμε για την αποτρεπτική ε, δράση της ε, αποστολής αυτής, ε, της επιχείρησης και αν μπορεί να παραμείνει, να είναι διαρκής η ισχύς και η αποτελεσματικότητά της. Και είναι πραγματικά στρατηγικής, στρατηγικού χαρακτήρα το ερώτημα του κατά πόσον μπορεί να παραμείνει αυτή η επιχείρηση. Οι στόχοι βέβαια εν μέρη ε, πληρώνονται γιατί εξακολουθεί να αναπτύσσεται η πειρατεία. Μήπως λοιπόν φτάνουμε στα όρια της επιχείρηση αυτή. Και όσο δεν εγγραφεί ε, σε πιο ε, ολοκληρωμένο πλαίσιο, με πιο ολοκληρωμένες δράσεις δηλαδή, θα είναι καταδικασμένη σε σχετική επιτυχία. Σε ό,τι αφορά τώρα το EUTM, Ποια είναι η χνηλασιμότητα, αν μπορώ να την αναφέρω έτσι, ότι αφορά την πρόσληψη προσωπικού που εκπαιδεύεται στην Ουγκάντα και στη συνέχεια αναπτύσσεται. Ε, μιλήσατε και για την αποστολή αλλά και για την προσωρινή κυβέρνηση ε, που αναλαμβάνει ουσιαστικά τα άτομα αυτά τα οποία προσλαμβάνονται πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πρόσληψη των σωστών ανθρώπων και στη συνέχεια τη σωστή ενσωμάτωσή τους για να μην μπουν σε άλλες ε, ομάδες ε, ισλαμικές ή, ισλαμιστικές ή οτιδήποτε άλλο. Πώς διασφαλίζεται λοιπόν την επιτυχία της διαδικασίας αυτής. Ε, είναι οι ερωτήσεις μου αυτές. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκουελχέρη. Grazie Presidente. Vorrei innanzitutto... Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον στρατηγό για την θαυμάσια παρουσίαση του θέματος, καθώς και για την προθυμία του να έρθει εδώ να μας μιλήσει. Είπε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα, όπως για παράδειγμα για την διάρθρωση της ε, εξωτερικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων. Τα όσα άκουσα συμβαδίζουν με τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Θα χρειαστούμε βέβαια μια δομή που να έχει την ικανότητα να συνδυάζει τις διάφορες πτυχές και διαστάσεις, διότι ακριβώς αυτό θέλουμε να μπορεί να κάνει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, δηλαδή να δημιουργεί συνέργειες από τις διάφορες προσεγγίσεις με συμμετοχή όλων των συνιστοσών. Είναι περίπλοκος τομέας αυτός. σιγά σιγά αρχίζει να αποκρισταλώνεται η δομή. Για παράδειγμα, πώς θα λειτουργεί η διοίκηση της επιχείρησης. Μένουν ακόμα πολλά να λεχθούν σχετικά. Και σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ των διαφόρων δομών, η CPD κτλ και του στρατιωτικού προσωπικού, του στρατιωτικού επιτελείου. Εάν δεν υπάρξει ένα ξεχωριστό όργανο, ένα ξεχωριστό διευθυντήριο, πώς θα λειτουργήσει την πράξη. Πώς θα γίνεται ο συντονισμός των διαφόρων δομών, αφού όλες έχουν διαφορετικές ευθύνες στρατηγικό σχεδιασμό από τη μια μεριά, πολιτικέ επιχειρήσει, δηλαδή μη στρατιωτικέ επιχειρήσει από την άλλη. Έχουν λοιπόν διαφορετικά καθήκοντα και το ερώτημα είναι πώς θα συντονίζονται. Για κάποιο διάστημα το Κοινοβούλιο συζητούσε τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού κέντρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γενικότερα, αυτό που ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο είναι ο χρονικός συντονισμός στρατιωτικών και μη επιχειρήσεων. Και όπως είπατε, και αυτή η συνολική προσέγγιση που είναι πολύ σημαντική στο πλαίσιο αυτό. Και πώς βλέπετε, πώς θεωρείτε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ομάδες μάχης σε επιχειρήσεις προστασίας πολιτών. Εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εκφράσατε κι εσείς και ο Πρόεδρος. Υπάρχει όντως μια απόσταση ανάμεσα στα όσα επέτυχε η Αταλάντη και στις προσδοκίες μας. Άρα πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η επιχείρηση Αταλάντη και να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιχειρήσεις μας και την αποδοτικότητά του τι επιχειρήσεις απέναντι και κατά τη πειρατεία. Μιλήσατε και για ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη τοπικών ηθαγενών δυνατοτήτων, ικανοτήτων. Τι εννοείται, τι θα μπορούσε να είναι το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος. Και ένα ερώτημα με εντονότερο πολιτικό χαρακτήρα που θα ήθελα να μου απαντήσετε αν είναι δυνατόν, καθώς επίσης να ακούσω και τις απόψεις και για τις επιχειρησιακές πτυχές του ίδιου θέματος. Εννοώ την αποστολή στο Κόσοβο. Σας ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για την έλευσή τους εδώ και για την επιθυμία τους και ε, προθυμία τους να περάσουν ε, κάποιο διάστημα μαζί μας για να συζητήσουμε σημαντικά θέματα και για την Επιτροπή μας αλλά και για όλη την Ευρώπη. Είπατε κάτι που με απασχολεί εδώ και χρόνια, δηλαδή αναφερθήκατε στο συντονισμό μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είδαμε και στον πόλεμο των Βαλκανίων και ιδιαίτερα στη Βοσνία είδαμε επικαλύψεις. Εγώ μάλιστα συμμετέσχα και σε μια επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Επιτροπή μας. Συναντηθήκαμε με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και το ξεκάθαρο μήνυμά τους ήταν να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε κάθε επικάλυψη γιατί είναι σπατάλη χρόνου και προσπαθειών. Εσείς αναφερθήκατε καμιά, και, στην, και είπατε μάλλον ότι ε, η πολιτική πτυχή καμιά φορά είναι αυτή που προκαλεί περισσότερα προβλήματα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτά που επιθυμούμε, τον συντονισμό δηλαδή μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης Μπορούμε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων που διαθέτουμε ή τα πολιτικά προβλήματα είναι τέτοιου μεγέθους που δεν μας επιτρέπουν να επιτύχουμε περισσότερα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο βέλτιστο της αποδόσεως ή νομίζετε ότι μπορεί να γίνει ακόμα πιο στενός συντονισμός ώστε να μην σπαταλώνται πόροι. Και ιδίω ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικός για την χώρα μου, τη Σουηδία, που δεν είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή μπορούν να συμμετάσχουν δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιες ε, αποστολές. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευρωπαϊκές δυνάμεις, χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό και ιδίως διότι εγώ διαβλέπω να αυξάνονται μάλλον οι ανάγκες για παρέμβασή μας προϊόντος του χρόνου και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και εκτός των οριών της ε, Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λέζινγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις εισαγωγικέ σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ και εσάς και τον Ζαν για τις ερωτήσεις σας. Θα δώσω κάπως πιο συγκεκριμένη διάσταση αφενός σε ό,τι αφορά την προέλευση των στρατιωτικών. Εγώ θέλω να ρωτήσω και σχετικά με την ηλικία, δηλαδή πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να εκπαιδευτούν και να χρησιμοποιηθούν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις παιδιά. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιχείρηση Αταλάντη ή τέλο πάντων την άμυνα κατά των πειρατών, θα ήθελα να μας δώσετε πιο ξεκάθαρους ορισμούς της επιτυχίας. Δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια για να θεωρηθεί μια τέτοια επιχείρηση επιτυχής. Επίσης, ερωτήσεις σχετικά με τις συνέργειες που αναφέρατε Υπάρχει από γερμανική, γαλλική και πολωνική πλευρά πρόταση για την δημιουργία ενός διαρκούς, ενός μόνιμου ε, επιτελείου στρατιωτικοπολιτικού. Τι γνώμη έχετε, ποια θα πρέπει να είναι η αριθμητική δύναμη καθώς και το κόστος που θα συνεπάγεται η δημιουργία ενός τέτοιου επιτελείου. Επίσης, ερώτηση σχετικά με την ένταξη του UNS στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων του UMS που είναι τμήμα του ΕΑΔ και εκεί θα πρέπει να συνεργάζονται χέρι με χέρι τα πράγματα αυτά στο μέλλον. Η ερώτησή μου είναι, μπορείτε να μας δώσετε μια ιδέα πώς βλέπετε την ανάπτυξη, την, πώς της τη συμμετοχή στην αναπτυξιακή βοήθεια τη δική σας και του UMS. Επίσης το EUMS συνεργάζεται από ό,τι είπε στενά με τον Οργανισμό Άμυνας. Τι μπορείτε να... Πώς, πού βρίσκονται τα προβλήματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα του μεταγωγικού αεροσκάφους ε, Airbus 400 ή του Γαριλαίου που έχουν κάνει και τόσο θόρυβο. Τέτοια σημαντικά προγράμματα, τέτοια σημαντικά εγχειρήματα έχουν νόημα για σας για το μέλλον, εφόσον προφανώς δεν ε, είναι η θέση οι υπεύθυνοι να μειώσουν το κόστος παρέλωσης της υποσχέσης τους. Η ε, κυρία και οι δικές μου ευχαριστίες βεβαίω και ζητώ, καθυστέρηση που, και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω αλλά τώρα με τις ερωτήσεις αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον τώρα συμφωνώ με τις ερωτήσεις της συναδέλφου μου σε ό,τι αφορά την πορεία της εξωτερικής δράσης τμήμα της οποίας είστε και εσείς 16 από τις 23 αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθαρά μη στρατιωτικού χαρακτήρα όμως στο επιτελείο σας, ποια είναι η αναλογία μεταξύ στρατιωτικού και μη στρατιωτικού προσωπικού. Γιατί μιλούμε εδώ για τις παρεμβάσεις σε πολιτικές επιχειρήσει, μη στρατιωτικές. Άρα χρειάζεται πολύ περισσότερο πολιτικό προσωπικό και όχι τόσο πολύ στρατιωτικό προσωπικό, παρόλο που ο ρόλος σα είναι σημαντικό, δεν το αμφισβητώ αυτό. Η αναλογία μου φαίνεται λίγο να γέρνει υπερβολικά υπέρ της πλευράς στρατιωτικών. και στο κέρας αφρική για παράδειγμα ε, όπου ε, απασχολείται θεωρητικό προσωπικό αλλά αυτές είναι οι αποστολές υπάρχουν κάποια στιγμή θα, θα σταματήσουν. Πώ πώς βλέπετε λοιπόν το μέλλον του επιτελείου σας αφού όπως είπα το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων μα θα είναι πολιτικού χαρακτήρα. Δεύτερο, μέσα στο ΝΑΤΟ ακούγονται σκέψει σχετικά με την κυβερνοάμυνα, ότι δηλαδή είναι σημαντική το βλέπετε ως μέρος του δικού σας έργου για το μέλλον. Εγώ βέβαια είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι σε αυτό, το λέω ήδη από τώρα. Πάλι για το ΝΑΤΟ, ορισμένοι εδώ σχεδιάζουν ενδεχομένως πολιτικές, δηλαδή μη στρατιωτικές ικανότητες του ίδιου του ΝΑΤΟ. Εγώ δεν το θεωρώ σκόπιμο αυτό. Εσείς που έχετε πολύ στενή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, πώς το βλέπετε. Τελευταίο τώρα. Επειδή εγώ είμαι Αυστριακή, δηλαδή από ουδέτερη χώρα, η ερώτησή μου είναι παρόμοια με τη συναδέλφου μου από την Σουηδία, που επίση είναι αδέσμευτη χώρα. Ποιο μπορεί να είναι ο ρόλος των ε, αδέσμευτων χωρών μέσα σε αυτήν την ευρωπαϊκή συνεργασία. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι σημαντικό, ειδικά στην ε, διαχείριση κρίσεων και ε, αποφυγή συγκρούσεων. Ο κ. Στάτσνη. πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούσαμε την παρουσίασή σας, γιατί όλοι οι συνάδελφοι χάρηκαν που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας για να, να συνεργαστείτε μαζί μας και να μας επιτρέψετε να συμμετέσχουμε στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνούμε και σε διαφορά αυτή τη συνολική προσέγγιση. Ήμουν και εγώ μεγάλος υπέρμαχος και χάρηκα που, υπάρξε, που υπήρξε ε, συνεργασία Βρετανών και Γάλλων, ιστορικών αντιπάλων. Ίσως η κατάσταση με την κρίση να προκάλεσε τη συνεργασία αυτή, αλλά ανεξάρτητα από το, το, τα αίτια της ε, συνεργασίας αυτής, συνέβη και είναι εξαιρετικό αυτό γιατί ακριβώς παρέχει αυτές τις συνεργασίες που χρειαζόμαστε και που αναφέρατε Μα ενώνει πιο πολύ και συνειδητοποιούμε ότι χρειαζόμαστε ο ένα τον άλλον. Ήμουν επίση μεγάλος υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωση ω υπερδύναμη, αλλά ξέρετε, συχνά είμαστε πολύ αδύναμοι. Χρειαζόμαστε τις δικές μας δομέ. Και αυτό στο παρελθόν προσπάθησαν να πετύχουν, για παράδειγμα, το RDU, το Rapid Deployment Units. Μιλάμε για αεροσκάφη για εξοικονόμηση, για παράδειγμα, πόρων. Θεωρείτε ότι υπάρχει προοπτική για μια καλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία. Με τη Γερμανία είμαστε, αντιπροσωπούμε ήδη ένα 80%. Αλλά νομίζω ότι θα χρειαστούν και οι άλλες χώρες. Αυτό το ένα σκέλος της ερώτησης και επίσης να ζητήσω τη γνώμη σας για το πώς βλέπετε την κατάσταση του Ιράκ και στο Αφγανιστάν σε 3 έως 5 χρόνια. Ευχαριστώ. General, thank you for your talk. σας ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω να σας θέσω. Η πρώτη είναι η εξής αν θα συμμετάχετε στην υπηρεσία εξωτερική δράσης, η πολιτική σας κατεύθυνση θα έρθετε από την υπότη εκπρόσωπο και όχι από τι εθνικέ κυβερνήσει στο μέλλον. Και δεύτερη ερώτηση. Μιλήσατε για τις περικοπέ στον προπολογισμό, το οποίο θα αναγκάσει τις εθνικέ κυβερνήσεις να συνεργαστούν. Και μιλήσατε για τη συμφωνία την Αγγλο-Γαλλική. Εγώ είμαι κατά, πολύ φοβάμαι, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι προδοσία των ε, εθνικών μας ε, συμφερόντων επικυριαρχίας. Χαίρομαι που υπήρξαν εξαιρετικά project, εξαιρετικά σχέδικα στρατιωτικής ε, ανάθεσης, αλλά νομίζω ότι αυτό το σύμφωνο παραπάει. Η δεν εμπιστεύονται τους Γάλλους ουσιαστικά και αυτό φαίνεται και σε ό,τι αφορά τα αεροπλανοφόρα. σε θέματα τεχνογλωσσίας και τεχνολογίας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι λάθος και αν πρόκειται μόνο για την περικοπή των εξόδων πραγματικά είναι καταδικαστέο αλλά ο σκοπός μας είναι πραγματικά ένας ενιαίος ευρωπαϊκός στρατός, ενιαίες ενόπλες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μία και μοναδική ατζέντα. Λοιπόν, θα βάλω τη σημαία μου του Ιταλική στην τσέπη για να μην μιλήσω καθόλου για τη χώρα μου. Βέβαια, σημειώνω με μεγάλη χαρά ότι δεν είπατε κάτι αντιγαλλικό. Εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη Γαλλία τουλάχιστον, από ό,τι φαίνεται. Ε, Δύο σύντομες ερωτήσεις ακόμη και θα ξαναδώσω το λόγο στο στρατηγό, ο κύριος Σκίνερ. Okay. Thank you Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Πίτερ Σκίνερ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον στρατηγό για την ε, παρουσίασή του. Δυστυχώς στο τέλος έφτασα, αλλά σίγουρα όλες οι προοπτικές μου φαίνονται πάρα πολύ ενθουσιώδεις. Ε, έρχομαι από μια περιφέρεια που χθε ή σήμερα ε, απελευθέρωσε δύο από τους δύο από τους ε, πειρατές που είχε ε, συλλάβει η Σομαλία. Καλό θα ήταν λοιπόν να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους ίδιους ομαλούς ώστε να μπορούν να αναφέρουν σε πέρας ε, και άλλα και ίδια τις επιχειρήσεις αυτές. Είπατε για, την, ε, για τον προπολογισμό. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ και για το διορισμό σας και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά και την παγκόσμια ασφάλεια και για το εμπόριο και για τα ταξίδια της μετακινήσεις ε, πράγματι δεν μπορούμε να περιμένουμε από τα πολιτικά σκάφη που είναι και πολλά αλλά πολύ μικρά και σίγουρα κάποιες φορές δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν ε, ε, τα, λίτρα που τους ζητούν γιατί φοβούνται και για τη ζωή τους και δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Αναγκόμες Στρατηγέ, πρώτα απ' όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη που δεν σας άκουσα προσωπικά, αλλά με ενημέρωσε ο βοηθός μου. Θα ήθελα να κάνω πάντως κάποια ερωτήματα. Εγώ είμαι μία από αυτούς που είμαι υπέρ της Γαλλοβρετανικής ε, Συμφωνίας ε, Συνέργειας, γιατί ό,τι και αν λένε κάποιοι, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα φέρει καρπούς ε, σε ό,τι αφορά το ότι θα ανοίξει προοπτικές για την ενισχυμένη χρήση των αμυντικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για τις επιπτώσεις ε, του νέου στρατηγικού δόγματος ε, του ΝΑΤΟ. Υπό την έννοια κυρίως ότι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού λέγεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος ε, εξειδίκευσης. Τα δύσκολα για τις ΗΠΑ και τα εύκολα το μη στρατιωτικό σκέλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ βέβαια εμείς πιστεύουμε και αντιλαμβανόμαστε βέβαια τη σημασία των μη στρατιωτικών δυνατοτήτων που έχουμε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε αυτές τις δυνατότητες μας να τις ε, θέσουμε στην υπηρεσία και του ΝΑΤΟ, αν όλα τα κρατημέλη βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν, αλλά δεν θα αφήσουμε τις δικές μας στρατιωτικές δυνατότητες κατά μέρο. Θα ήθελα επίσης να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Όπως φαίνεται, Υπάρχει μια νέα ε, συμφωνία για την πυρηνική θέση, την θέση ότι αφορά ε, τα πυρηνικά. Ακούσαμε διάφορε απόψει από διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε και τη νέα πυρηνικό δόγμα των, ε, και την πυρηνική στάση των ΙΠΑ Πιστεύετε ότι τελικά θα υπάρξει κάτι καινούριο στο ΝΑΤΟ ή όχι. Και τελικά τι είναι αυτό, θετικό αρνητικό. Για μένα είναι αρνητικό γιατί δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη, ε, ούτε το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να ηγηθεί ενό πολύ σημαντικού ζητήματος ε, πολέμηση αποτελεσματική της διάδοσης. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Στρατηγία σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα μετέθεσαν. Θα προσπαθήσω να συνδυάσω ορισμένα από αυτά. Και για τα διαφορετικά θα διατρέξω τον κατάλογο. Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση Αταλάντη και τι μπορούμε παραπάνω να κάνουμε, νομίζω το έθεσαν τουλάχιστον δύο βουλευτές, εκ των οποίων ένας ήταν ο πρόεδρος της υποεπιτροπής σας. και τι θα πει αποτελεσματικό, με ρώτησε κάποιος. Θα ξεκινήσω με τη δήλωση ενός από τους βουλευτές. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς, να μην κάνουμε τίποτα. Να αφήσουμε τους πειρατές ε, να δρούν ανενόχλητοι, ε, θα ανεβούν οι τιμές γιατί θα πιάσουν ε, πολλά, πιο, πολύ περισσότερα εμπορικά πλοία, η βιομηχανία θα έχει προβλήματα και ούτω καθεξής. Επομένως είναι και συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει κάτι. Όχι όμως μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και ε, το συμφέρον της ε, Κίνας, της Ινδίας, των ΙΠΑ. όλοι δηλαδή ενδιαφέρονται, όλοι έχουν συμφέρον να καταπολεμηθεί η πειρατεία. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκεί υπό το καλύτερο δυνατό πλαίσιο. Γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες δυνατότητες κράτη-μέλη, αλλά και κράτη-μέλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή την επιχείρηση Αταλάντη, την Ευρωπαϊκή. Γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί οι κανόνες εμπλοκής μας και το νομικό μας πλαίσιο είναι, γέννη, είναι το πιο ενδιαφέρον. Και γιατί έχουμε και περισσότερες δυνατότητες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε συμφωνίες με την Κένια, με τις Αιγέλες έχουμε συμφωνία και ελπίζουμε να έχουμε και με άλλες χώρες συμφωνία. Έτσι θα μπορέσουμε να καταδιώκουμε τους πειρατές στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά και κανείς δεν θέλει τους πειρατές στη δική του χώρα ε, και καλό να τους συγκεντρώσουμε σε μια περιοχή. Γιατί λοιπόν έχουμε συμφωνίες και άλλοι θέλουν ή δεν θέλουν να τις έχουν αυτές. Όχι γιατί, ε, μάλλον γιατί δεν είμαστε μόνο στρατιωτικός παίκτη, αλλά και εμπορικός εταίρος γενικώ. Και θέλουν να κάνουν δουλειές μαζί μας, έχουν επιχειρηματική σχέση μαζί μας πολλές χώρες. Και έτσι και το στρατιωτικό σκέλος ενισχύεται και γίνεται πιο αποτελεσματικό. Είναι σαφές ότι αν συνεχίσουμε μόνο με δράσεις καταπολέμησης της πειρατείας, αυτό δεν θα είναι αρκετό. Τελικά ε, χρειαζόμαστε περισσότερα πλοία γιατί οι πειρατέ ε, μαθαίνουν, ξέρετε. Δεν μαθαίνουμε μόνο εμείς και γίνονται πιο έξυπνοι. Πρέπει λοιπόν ε, να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του κακού που βρίσκεται στη Σομαλία, στην ξηρά η κυβέρνηση που υπάρχει εκεί, που δεν είναι κυβέρνηση ουσιαστικά, αυτή που υποστηρίζουμε είναι η λεγόμενη TFG, Transformation Federal Government, ένα έδος ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αλλά όσο δεν υπάρχει κάτι άλλο θα συνεχίσουμε ε, τις δράσεις πολέμηση της πειρατείας. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα στη Σομαλία, αλλά όχι όμως μόνο στη Σομαλία, γιατί θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και αποφελές ε, να έχουν καλύτερες δυνατότητες καταπολέμησης της πειρατείας και οι άλλες χώρες της περιοχής και έπειτα έχουμε ένα ε, σύστημα για να έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Δημιουργία εκτοφυλακής, ναυτικής ε, δυνατότητας, δηλαδή για την καταπολέμηση πειρατείας από την ίδια τη χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα ως ιδέα να το υποστηρίξω. Και βέβαια, στο πλαίσιο της ε, υπηρεσίες εξωτερικής δράσης που είναι υπό ανάπτυξη δεν υπάρχει ακόμη, δεν είναι επιχειρησιακή. Με ό,τι έχουμε τέλος πάντων στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε ιδέες ε, για να τις υποστηρίξουμε και σίγουρα υπάρχει συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι πολύ σημαντικός εταίρος. Όχι μόνο ε, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά γενικώ ένας πολύ σημαντικός εταίρος Βέβαια σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα δεν είναι στρατιωτικού χαρακτήρα. Αλλά ναι, πράγματι έχω και κάποιες ιδέες για το τι μπορεί να κάνει το στρατιωτικό σκέλος. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την πλοήγηση, ε, στο τι μπορεί να κάνει το ναυτικό, τι μπορεί να κάνει το ναυτικό και ε, η πολιτική πλευρά, το μη στρατιωτικό σκέλος, αλλά Υπάρχουν και άλλα μέσα που έχει στη διάθεσή τη η Κομισιόν και να και στην Επιτροπή να δει κατά πόσον θέλει να τα χρησιμοποιήσει ή όχι. Εγώ πάντως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να συζητάμε μεταξύ μα και βέβαια να δούμε πώς μπορούμε να ε, συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί κάποιες φορές η αναπτυξιακή βοήθεια είναι εντελώ άχρηστη αν δεν υπάρχει ασφάλεια. Και κάποιες φορές δεν είναι καν χρήσιμο να πάει κανείς ε, ως στρατός και να δημιουργήσει την ασφάλεια αν δεν υπάρχει κάποια δράση ανάπτυξη στη χώρα από κάποια άλλη πλευρά. Η πατή πρόσωπος έχει και την αρμοδιότητα του συντονισμού. Ο συντονισμός δεν είναι όμως ε, ποιος ε, είναι πάνω από τον άλλον. Ε, ουσιαστικά εξηγείς τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να κάνει ο άλλος, ώστε τελικά να υπάρχει μια συνεργασία και να λαμβάνονται κοινά οι αποφάσεις για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, που υπάρχει όταν υπάρχει συντονισμός. Τώρα, τι ακριβώς θα συμβεί. Φυσικά εγώ δίνω τις συγκεκριμένες μου ιδέες για το πώς μπορούν να επιτευχθούν κάποια πράγματα και ένα από τα ερωτήματα ε, ήταν αυτό ακριβώς, ε, πού αναφέρομαι και πώς αναφέρομαι. Εγώ δίνω στατητικές συμβουλές μέσω της ιεραρχίας, μάλλον όχι μέσω της ιεραρχίας, δίνω τις στρατιωτικές μου συμβουλές στην ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο που έχει ίδια την ευθύνη του συντονισμού, να έχουμε λοιπόν συντονισμένες ιδέες και αυτό μπορώ να το κάνω απευθείας, άμεσα, μέσω του συντονισμένου μηχανισμού που έχουμε. Το CMPD, το Κέντρο Διαχείρισης ε, Κρίσεων ε, και στον της κυρίας Κλωτ Φρανς ε, είναι πολύ σημαντικό για το στρατηγικό σχεδιασμό στρατιωτικό, πολιτικο-στρατιωτικό. Και εγώ λοιπόν για το τελευταίο σκέλος αναφέρομαι σε αυτή. Δεν είναι το αφεντικό μου βέβαια. Είναι όπως στο πλαίσιο του στρατιωτικού επιτελείου. Έχεις ε, το στρατηγικό τμήμα, το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τις τρέχουσες επιχειρήσεις. Δεν είναι, είναι κανείς προϊστάμενος του άλλου. Το θέμα είναι πού βρίσκεται η διαδικασία σε κάθε περίπτωση. Στο μακροχρόνιο προγραμματισμό, αν είσαι σε αρμόδιος ή άλλοι σου δίνουν input, αλλά όλοι ουσιαστικά αναφέρουμε στον ίδιο διοίκηση. Εγώ είμαι γενικός διευθυντής του στρατιωτικού επιτελείου αυτή τη στιγμή. Εμείς ε, με τους άλλους συνεργάτες μου επικοινωνούμε, προσπαθούμε να καταλήξουμε ε, στον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό. Συζητούμε με την είπατε πρόσωπο που είναι πολύ ικανοποιημένη. Το ίδιο όμως είμαι και εγώ γιατί και είπατε εκπρόσωπο μπορεί να συντονίσει πολύ περισσότερους από αυτούς που μπορούσαμε εμείς πριν από λίγα χρόνια. Και σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική αποστολή, το EUTM επίσης έχω άμεση ε, εμπλοκή. Ε, αναλάβαμε κάποιο ρόλο, κάποιες αρμοδιότητες στην πρόσληψη και στην εκπαίδευση. Βέβαια αυτή ουσιαστικά ε, την έχει αναλάβει η κυβέρνηση, TFG, αλλά βοηθά πολύ ε, και Βοηθούν και οι ΙΠΑ, ε, μεταξύ άλλων, είναι πολύ σημαντικός ε, εταίρος. Μετά έρχονται σε εμά. Γίνεται και επιλογή από πλευράς μας. Δηλαδή όλους τους ε, εκπαιδευόμενους τους βλέπουμε. Ελέγχουμε, τους ελέγχουμε. as well. Ε, Βλέπουμε την ηλικία τους για να μην είναι παιδιά και γενικώ προσπαθούμε να τα ταυτοποιούμε όλα τα άτομα, να υπάρχει αναγνώριση, ε, ώστε για παράδειγμα χάρη και την πληρωμή να την παίρνουν οι στρατιώτες και όχι κάποιοι άλλοι. οι οποίοι μισθοί αυτοί καταβάλλονται από τη ΣΥΠΑ. Λοιπόν, ε, δεν είναι δική μου ευθύνη. Είναι εκτός δική μου ευθύνη, αλλά ε, κάνουμε κι εμεί ε, πολύ εξονυχιστικό έλεγχο. Και θέλουμε να δούμε και όταν ενταχθούν στην TFG, στην Transformation Federal Government, θέλουμε να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. η αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ναϊρόμπι συχνά έχει επαφές λοιπόν με αυτή την κυβέρνηση και ελέγχει τα πράγματα. Έπειτα, σε ό,τι αφορά την ΕΕΦ, την, εξωτερική, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, είναι μια ερώτηση που μου τίθεται συχνά πώς αυτή η συνεργασία ε, στρατιωτικού με στρατιωτικού σκέλους ε, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Κατ' με όταν υπάρχει κρίση καλούνται στο ίδιο τραπέζι όλοι. Ε, με πρόεδρο βέβαια την είπατε εκπρόσωπο, ενώ αν δεν είναι αυτή θα είναι γενικό γραμματέα που θα προεδρεύει. Πάντω είπατε εκπρόσωπο συνήθω θέλει να είναι εκεί και προσπαθούμε να είναι εκεί τι περισσότερε φορέ. Στο Πακιστάν, παραδείγματο χάρη, έγινε αυτό. Όλοι λοιπόν οι σημαντικοί παίκτε κάθονται στο ίδιο τραπέζι και το στρατιωτικό σκέλος, η SMTPD και, το, και άτομα από την Κομισιόν. Και έτσι γίνεται μια συζήτηση, ποιο είναι το πρόβλημα, θα πρέπει να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν ναι, ποιο θα πρέπει να είναι ο στόχο, και αφού βρούμε το στόχο, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ε, θα πούμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε το στρατιωτικό σκέλος, άρα εγώ δεν συμμετέχω πάντοτε σε όλες αυτές. Υπάρχει όμως κάποιες φορές η απόφαση ότι μπορεί ενδεχόμενος να χρησιμοποιείται το στρατιωτικό σκέλος. Βέβαια, είπατε εκπρόσωπος δεν είναι αυτή που αναλαμβάνει πάντοτε το συντονισμό, γιατί καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί πάντως ε, που είναι υπό την αιγίδα της ε, ξέρουμε ότι αναπτύσσει και τις διαδικασίες και όταν υπάρχει ε, συμμετοχή του αγροτικού σκέλου, ε, υπάρχει υπόσχεση ότι εγώ πάντοτε θα συμμετέχω από την αρχή. Και θα δούμε ποιο στρατιωτικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί, εάν χρειαστεί. Τώρα, σε κατώτερο επίπεδο, πώς λειτουργεί. Έχουμε το CMPD που έχει τον συντονιστικό ρόλο για, τις, για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αυτό θα προχωρήσει, θα για να δούμε πώς θα γίνει ο συντονισμός. Υπάρχει ένα επόμενο επίπεδο, βέβαια, προς τα κάτω που θα είναι το επιχειρησιακό επιτελείο. Κάποια στιγμή του χρόνου θα ξαναγίνει συζήτηση. Αυτό αναμένω. Διάβασα την εκθεσή σας. Για δεύτερη φορά εσείς ζητείτε να το επανεξετάσουμε. Βεβαίως το επανεξετάζουμε και θα το επανεξετάσουμε του χρόνου, διότι φαίνεται λογικό Ωστόσο να αναμείνουμε πρώτα να αναπτυχθεί η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων όπου θα γίνει ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση αυτής της συνολικής ε, προσέγγισης και μετά να αρχίσουμε τις συζητήσεις σχετικά με το τι να κάνουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσεγγίσει κανείς το θέμα. Σας ευχαριστούμε για τις ε, προτάσεις σας, για την σύστασή σας να γίνει δηλαδή ένα διαρκές επιτελείο και εκεί να συστεγαστούν ε, πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εγώ βέβαια θα συμβάλλω με την άποψή μου. Υπάρχουν σαφή, ε, συγγνώμη, σαφή πλεονεκτήματα του τρέχοντος συστήματος, του σημερινού συστήματος, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Είτε για παράδειγμα τα πέντε εθνικά ε, επιτελεία ή η δική μου επιχειρησιακή ικανότητα Υπάρχουν διάφορε δυνατότητε. Όλε αυτέ έχουν βέβαια και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά όλα μαζί σε συζήτηση βέβαια και με του άλλου εταίρου μα γιατί εγώ μπορώ να σα δώσω την άποψή μου, αλλά είναι πιο ευγενέ νομίζω να περιμένω μέχρι του χρόνου και να υποβάλω ένα έγγραφο το οποίο ασφαλώς θα συνταχθεί ε, για το θέμα δηλαδή πώς μπορεί να γίνει καλύτερος ο συντονισμός. Ασφαλώς και είναι σημαντικό να εξεταστεί. Μετά και πάντοτε για την συνολική προσέγγιση για τις ε, μάχημες ομάδες. Η, η ίδια η έννοια των μάχημων ομάδων, εκεί λαμβάνουμε υπόψη ορισμένα σενάρια σχετικά με την υποστήριξη, διότι μέσα στην έννοια της ε, battle group, της μάχημης ομάδας, είναι εάν υπάρξει μια τεράστια ε, ανθρωπιστική καταστροφή, μπορούμε τότε να χρησιμοποιήσουμε τις μάχημες ομάδες. Και πάντοτε ο στρατιωτικό σκέλος θα είναι σε υποστήριξη, ποτέ δεν θα έχει τον ηγετικό ρόλο. Ποτέ δεν θα πει ε, το στρατιωτικό σκέλος πώς θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο. Αλλά είναι καλύτερα βέβαια να συζητούμε για να ε, τα κάνουμε με ασφαλή τρόπο αν δεν υπάρχει ασφάλεια, εκεί μπορεί να βοηθήσει ο στρατό σε μια μεγάλη ας πούμε, ανθρωπιστική καταστροφή για την διασφάλιση τη ασφάλεια. Αλλά οι μάχημε ομάδε δεν είναι φτιαγμένε για να ε, αντιμετωπίζουν καταστροφέ και δεν πρόκειται να γίνει κιόλα, διότι οι χώρε μέλη θέλουν τι μάχημε ομάδε να μπορούν να δράσουν ε, ταχύτατα ε, σε στρατιωτικές περιστάσεις. Έχουν λοιπόν και την μάχημη ικανότητα. Ορισμένες από τις μονάδες αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανθρωπιστική βοήθεια. Ένας φαντάρος του πεζικού μπορεί να βοηθήσει να κουβαλήσει ας πούμε ε, ανθρώπους που είναι ανίκανοι να κινηθούν μόνοι τους ή να βοηθήσει να φτιαχτούν φράγματα με ε, τσουβάλια άμμο και ασφαλώς βέβαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δυνάμεις αυτές και για ε, ιατρική υποστήριξη για παράδειγμα κτλ. Η απάντησή μου προκειμένου πάντως θα είναι ότι εάν σχετίζεται, εάν είναι τμήμα δηλαδή μιας συνολικής προσέγγισης, ασφαλώς αυτό θα γίνεται, θα γίνεται πάντοτε σε συντονισμό με τις άλλες προσπάθειες και όχι ε, με ηγετικό ρόλο του ε, σταθερικού ε, σκέλους. Γιατί να τα λάβει απάντησα ήδη. Τώρα, η αποστολή στο Κόσοβο. Μπορώ να σας πω την άποψή μου, αλλά δεν έχω εντολή και δεν υπάρχει στρατιωτική αποστολή στο Κόσοβο. Για μένα το πιο ενδιαφέρον και σημαντικό είναι να έχουμε, ότι έχουμε αν κοινού πόρου εκεί, μοιραζόμαστε τους πόρου, και αυτό με φαίνει στη συνεργασία στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Εάν πρόκειται τώρα για συνεργασία Ευρωπαϊκή στη Βοσνία Ζεγοβίνη, αυτή είναι εξαιρετική είναι πραγματικά άριστη. Είναι Βερολίνο συν. Δεν νομίζω θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική. Αυτό θα απαντήσω και είναι ήδη εξαιρετικά επιτυχημένη ως έχει. Θα έχουμε και άλλη επιχείρηση Βερολίνου συν. Αυτό δεν είναι δική μου απόφαση βέβαια. Είναι απόφαση ε, των πολιτικών ηγετών και όλοι γνωρίζουμε ότι ίσως να υπάρξουν δυσκολίες σχετικά με μια επόμενη ε, αποστολή Berlin Plus. Ο, ο, ε, ανώτατος συμμαχικός διοικητής δυνάμεων στην Ευρώπη είναι αυτός που είναι διοικητής εδώ των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Αυτός δηλαδή χρησιμοποιεί το επιτελείο του στο επίπεδό του και έχει και βέβαια και υποστήριξη του ε, ΝΑΤΟ από το αρχηγείο της Νέα Πόλεως, της Νάπολη ε, στη Βοσνία και βεβαίω γίνεται και ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Ακριβώ επειδή είναι επιχείρηση Βερολίνου ΣΥΝ. Εφόσον λάβει ευρύτερο χαρακτήρα, τότε η συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται δυσχερέστερη, γιατί αν δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό το Βερολίνο ΣΥΝ, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Επίση. για Τέλο πάντων, θα δούμε για το άλλο θέμα που μου θέσατε, εάν θα ε, μπορέσουμε να δράσουμε ε, ναι, για την Αταλάντη, όπω είπαμε, τα είπα. Για την συνεργασία στα ιδιωτικού και μη στρατιωτικού τομέα. Ε, νομίζω τα είπα αυτά αρκετά, αν σας ικανοποιήσει η αποτίμηση μου για αυτό το περίφημο Σιβ Μιλ, θα υποβάλουμε προτάσεις. Δεν μπορώ όμως να ε, προβλέψω από τώρα ποια θα είναι η αριθμητική δύναμη του προσωπικού. Διότι αυτό θα εξαρτηθεί από την ε, κοινή συμφωνία. Αν αρχίσω να λέω νούμερα τώρα, ε, νομίζω θα είναι πολύ πρόωρο. Αυτό άλλωστε θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή η, η άποψή μου θα πρέπει να υποβληθεί πρώτα μέσα στην ε, στι στρατιωτικέ δομέ, στι ε, ιεραρχικέ μου δομέ και μετά. Αλλά τέλο πάντων θα το συζητήσουμε αυτό. Ο, ο ρόλος της EUMS για την αναπτυξιακή βοήθεια. Έχω κάτι πει σχετικά ήδη. Καμιά φορά υπάρχουν σοβαροί λόγοι η αναπτυξιακή βοήθεια να μην συνδυάζεται με στρατιωτική παρουσία. Και γιατί, διότι η άνθρωποι που εργάζονται στην ανθρωπιστική ή στην αναπτυξιακή μάλλον βοήθεια και που είναι συχνά μη κρατικέ οργανώσεις έχουν συχνά προστασία, χαίρουν προστασία, ακριβώ από το γεγονό ότι δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικού. Και οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν σε πάρα πολύ δύσκολε ε, ε, περιοχές ε, χωρίς προστασία και το κάνουν αυτό επειδή φαίνονται, ε, έχουν την εικόνα του ουδετέρου ασφαλώς εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και έχω απόλυτο σεβασμό για όσου τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε όμω και πολλά παραδείγματα όπου δίνεται αναπτυξιακή βοήθεια χωρί καμία περιφερειακή ασφάλεια και εξαφανίζεται κάπου η αναπτυξιακή βοήθεια χωρί κανένα ε, αυτό αποτέλεσμα. Και τότε βέβαια τίθεται το ερώτημα ποιο μπορεί να είναι ο ρόλο του στρατιωτικού τομέα εκείνη τη στιγμή. Και γνωρίζουμε ότι έχουμε και πολλά παραδείγματα όπου μη κρατικοί οργανισμοί αρχικά δεν ήθελαν να συνεργαστούν με τι στρατιωτικέ αρχέ ακριβώ λόγω του πρώτου επιχειρήματο που σα έδωσα, τώρα έρχονται και ζητούν την υποστήριξη του στρατού. Η Αταλάντη, για παράδειγμα, ο λόγο για τον οποίο αρχίσαμε ήταν ότι το World Food Program μα ζήτησε να του υποστηρίξουμε και να συνοδεύουμε τα πλοία του, τι νιοπομπές του. Το World Food Program επειδή τα γνωρίζω και από την προηγούμενη δουλειά μου, το World Food Program στο Αφγανιστάν δεν ήθελε στην αρχή την ε, υποστήριξή μας. Τώρα συνοδεύουμε ε, τις εφόδιο τους στο Αφγανιστάν και είναι και πολύ ευχαριστημένοι και δεν έχουν αλλάξει άποψη. Υπάρχουν και άλλα πολλά σχετικά παραδείγματα. Τώρα, σχετικά με το Αφγανιστάν, δεν έχω βέβαια ευθύνη, ε, δεν φέρω ευθύνη για τα θέματα αυτά, διότι αυτά είναι civilian inputs. Εκεί εγώ δεν έχω, όπως είπα, κανένα τομή ευθύνη, αλλά σε προηγούμενες θέσεις που κατήχα και επειδή εξακολουθώ να παρακολουθώ το τι γίνεται εκεί, αποδεικνύεται ότι ο μόνος τρόπος να επιτύχουν οι επιχειρήσεις να σχεδιάζει κανείς ταυτόχρονα και τα δύο σκέλη και το πολιτικό και το στρατιωτικό της επιχείρησης και όχι μόνο στρατιωτικό και μετά να σκεφτούμε τι θα γίνει με την ανάπτυξη της ε, χώρας. Εγώ μπορώ να προβλέψω ότι σε πολλές περιπτώσεις τον ηγετικό ρόλο θα αναλαμβάνουν οι πολίτες, δηλαδή οι μη στρατιωτικοί και μετά θα, ρωτήσουν, θα ρωτήσετε ποιος θα είναι ο δικός μας ρόλος. Το Πακιστάν ωστόσο είναι καλό παράδειγμα. Συνέβη ανθρωπιστική καταστροφή, για πολλούς λόγους δεν ήταν σκόπιμη στρατιωτική παρουσία, αλλά τουλάχιστον μπορέσαμε να, μπόρεσα να προσφέρω την, τις μεταφορικές ικανότητες. Και η Κομισιόν είπε ευτυχώς, διότι δεν είχε επαρκείς μεταφορικές ικανότητες και χρησιμοποίησε τις δικές μας. Και αυτό, αυτός είναι ένας καλός τρόπος συνεργασίας. Και ήταν τελείως ανόητο που κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να συμβεί εδώ και λίγα χρόνια, πριν από λίγα χρόνια δηλαδή. ανάπτυξη ικανοτήτων. Δεν μπορώ να διαβάσω ακριβώ τη σημειώση μου. Τι με ρωτήσατε ακριβώ τελευταία σα ερώτηση, κυρία Λέσινγκ. Α, το κόστος του Airbus 400. Μπορώ να σας δώσω πολλά μη στρατιωτικά προγράμματα που ξεκινούν και μετά εγκαταλείπονται διότι είναι εξαιρετικά δαπανηρά. Για μένα λοιπόν αυτό δεν είναι λόγος. Αλλά εσείς βέβαια είστε βουλευτές και ως βουλευτές είστε υποχρεωμένοι να επιμένετε στην τήρηση των δημοσιονομικών πλαισίων. Αυτό που βλέπω ωστόσο εγώ είναι μία από τις μεγάλες ελλείψεις, ειδικά στην Ευρώπη, ότι εξαρτώμαστε τόσο πολύ από άλλους. Για παράδειγμα, ε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν σημαντική μεταφορική ικανότητα ή ε, μισθώνουμε ή ναυλώνουμε μεγάλα ε, μεταγωγικά αεροσκάφη αντόνοφα από την Ουκρανία, αλλά μας κοστίζουν πολλά. Δεν έχουμε λοιπόν μεταγωγική ικανότητα για διαφόρους λόγους. Ο μόνος τρόπος λοιπόν που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό είναι να έχουμε κοινού τύπους ο αριθμός και κοινά αεροσκάφη. Ο αριθμός δηλαδή των αεροσκαφών που απαιτείται δεν μπορεί να τον επομιστεί μονάχα μια χώρα. Το α400 μη θα είναι τμήμα αυτού του ε, project της ADF για την EDA έχει βέβαια ε, θετικό ρόλο, είναι, είναι, είναι κάτι που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι όμως ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. διότι αν γίνει η ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πρέπει να συμφωνήσουν όλε οι χώρε μέλη με την χρήση της ε, ικανότητα αυτή. και μόνο μία χώρα, και μία μόνο χώρα δηλαδή, θα μπορούσε ε, να την ακυρώσει, να προβάλλει βέτο δηλαδή. Άρα δεν είναι σωστό τρόπο αυτό. Γι' αυτό και από την ερώτηση, στοχεύουμε σε <coughs> στρατιωτικές δυνάμεις της Ένωσης, αυτό σημαίνει ή θα σήμαινε ότι πάμε να φτιάξουμε μια ικανότητα την οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Αυτό που χρειάζεται είναι οι χώρε μέλη να δημιουργήσουν ικανότητε και υποπελίτε που εάν θέλουν κάποτε να τι χρησιμοποιήσουν. Εφόσον αποφασίσουν μια, εγκρίνουν μια αποστολή, τότε ελπίζω να έχουν και τι ικανότητε. Εάν όμως η επιχείρηση τοποθετηθεί σε ύψο στο επίπεδο ενό άλλου διεθνού φόρουμ, τότε να μπορούν να συμμετάσχουν οι χώρε. Τώρα, το Airbus 400, το EATC είναι επίση ένα θαυμάσιο παράδειγμα ε, συνεργασία ή συντονισμού μάλλον. Και βλέπω μάλιστα και την Βρετανογαλλική συνεργασία με τον ίδιο τρόπο. Η δική μου ερώτηση θα είναι τι είναι καλύτερο, να μην υπάρχει καθόλου ικανότητα ή να υπάρχει κοινή ικανότητα. Εάν μου πείτε θέλω δική μου ικανότητα και θα τα πληρώσω μόνος μου, θαυμάσια. Αλλά δεν θα λύσει το οικονομικό πρόβλημα του Ηνωμένου Βασιλείου κάτι τέτοιο. Τα καλά νέα λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και νομίζω και όλες οι χώρες μέλη και διερωτώ με γιατί αναστατώνονται τόσο πολύ ορισμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και θεωρούν ότι δεν είναι ευρωπαϊκό. Ανησυχήσατε για την Ολλανδογερμανική συνεργασία στα, στο επιτελείο ή για τη βαλτική συνεργασία των χωρών της Βαλτικής. Δηλαδή, όχι. Αυτά είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι οι χώρες μέλη μόνο εφόσον συνεργαστούν μπορούν να δημιουργήσουν κοινέ ικανότητε και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει το ρόλο του διευκολυντή διότι βάζουν κάτω όλες τις απαιτήσεις τους χώρες μέλη και εμείς κάνουμε το συντονισμό. Λέμε εσύ και εσύ και εσύ έχει αυτή την απέτηση, α συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε την ικανότητα. Αυτό είναι ο στόχο μας. Μάλιστα. Ίδιο μες 200. Ναι, αν είναι καλή αναλογία. Να σας δώσω λίγα παραδείγματα. είναι 299 στην πραγματικότητα. Έχουμε 199 στρατιωτικούς. Ανάμεσα σε περίπου 30.000 πολίτες. Δεν λέω ότι είμαι πολύ ψηλός, δεν λέω ότι είμαι και πολύ κοντός. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το μικρό μπορεί να είναι και αποτελεσματικό. Ορισμένοι εκτός της αίθουσας σας έχουν πει ότι είναι υπερβολικά στατιωτικοί. Μα εγώ λέω είναι 7 στατιωτικοί και όλοι οι υπόλοιποι είναι πολιτικό προσωπικό. Ίσως φαινόμαστε πιο πολύ επειδή ε, πάμε στη δουλειά ένστολη, φορώντας τη στολή δηλαδή. Εγώ πάντως είμαι ικανοποιημένος από τους αριθμούς αλλά είμαι και ικανοποιημένο και από τη συνεργασία με του άλλου. Τώρα, κυβέρνω άμυνα, θα είμαι σύντομο. Δεν έχουν ληφθεί ακόμα επισήμως αποφάσει. αλλά ε, μπορώ να προβλέψω ότι η πολιτική αυτή θα κριθεί ω πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. αλλά ο στρατό δεν θα έχει ηγετικό ρόλο καθόλου στο θέμα αυτό. Ο στρατός θα παραμείνει σε επαφή, διότι έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε τα δικά μας συστήματα απέναντι σε οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση. Αλλά δεν βλέπω να διαγράφονται κάποιες εξελίξεις που να δώσουν στις ενόπλες δυνάμεις άλλο ρόλο, εκτός από το να προστατεύσουν τα δικά τους συστήματα. Τώρα έχω και ορισμένες άλλες ερωτήσεις σχετικά με το ΝΑΤΟ, την ε, δημιουργία πολιτικής, δηλαδή μη στρατιωτικής ικανότητας. Γνωρίζετε ότι είναι πολύ περιορισμένη. Το ΝΑΤΟ δεν αναπτύσσει δικές του πολιτικές ικανότητες ή όργανα. Το μόνο που κάνουν, και αυτό είναι σημαντικό βήμα κατά τη γνώμη μου, σε κάθε ε, στρατηγείο βάζουν και ένα πυρήνα ένα πυρήνα πολιτικής συνεργασίας. Υπάρχει αυτό που λέμε σύμικ που είναι ωστόσο τμήμα της επιχείρησης. Δηλαδή αν θέλετε να είναι αποτελεσματική η στρατιωτική επιχείρηση, αλλά θέλετε ταυτόχρονα να κερδίσετε την εμπιστοσύνη και ε, την υποστήριξη των πολιτών, χρειάζεται και αυτή η ΣΥΜΙΚ ε, ε, πτυχή. Το ΝΑΤΟ τώρα, όπως και εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται πολύ περισσότερο από αυτό. Το ΝΑΤΟ αντιλαμβάνεται ότι η επιχειρήση του θα είναι επιτυχής εφόσον συνεργαστεί και με πολλούς άλλους civilian players, όχι μόνο του ΝΑΤΟ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι κάποιος από τους ε, εταίρους, η παίκτες αυτούς, αλλά άλλοι, άλλοι μπορεί να είναι μη κρατικοί οργανισμοί ή μπορεί να είναι οι τοπικές αρχές. Άρα χρειάζεται μια συντονισμένη ικανότητα, η οποία δεν υπήρχε πριν, για να επιτευχθούν αυτά, για να είναι αποτελεσματικέ επιχειρήσει. Το έχουν αποφασίσει να αναπτύξουν την ικανότητα αυτή και αυτό είναι καλό για δύο λόγου. Αφενό, διότι είναι εφικτό Αφετέρου και ίσως πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει πάντοτε ένας επικεφαλής ο οποίος αναλαμβάνει την, ε, τον συντονισμό αυτών του, του πολιτικού δηλαδή τομέα. Κάθε φορά που ο στρατιωτικός διοικητής φαίνεται να λησμονεί την ανάγκη να λάμβει υπόψη του και τις ε, απόψεις αυτές. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα και να υπάρχει ένας τέτοιο γενικός σύμβουλο σε όλα τα επίπεδα. Δεν το είχαμε αυτό μέχρι τώρα στην οτροπία μας. Διότι βάζουμε κάτω τα ε, ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και βλέπουμε ότι το ζητάνε αυτό και εγώ βλέπω ήδη αποτελέσματα διότι το πρόσωπο αυτό μπαίνει μέσα στην διαδικασία λήψη απόφαση, σηκώνει το χέρι του και λέει αν θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, θα τα πει κύριε Δικητάν, πως ξεχνάτε και το υπόλοιπο 50% του κόσμου, του κοινού, ε, στην χώρα που γίνεται επιχείρηση. Αυτό είναι σημαντικό, διότι ορισμένες φορές τα λησμονούσαμε αυτά τα πράγματα. Μιλούσαμε μοναχά στους επικεφαλείς των διαφόρων κλάν, των μεγάλων ε, ομάδων ή οικογενειών. Είναι καλύτερα να μιλούμε και στις μανάδες των γιών που είναι οι ταραξίες. Τώρα, εφόσον κανείς είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κοινή ευθύνη βεβαίως για την οικονομία, για την κοινή αγορά, για κοινή ασφάλεια. Αυτό περιλαμβάνει και την ασφάλεια και άμυνα και ο ρόλος που αναλαμβάνει η χώρα σας εν προκειμένου είναι πολύ θετικός και τον υποστηρίζω. Δεν αφαιρεί κανένας είδους κυριαρχία ή επιλογές. Ε, και μιλώ βέβαια για τις αδέσμευτες χώρες. Μας μένουν μεταξύ 5 και 7 λεπτών ακόμα στρατηγέ μου, άρα ας προσπαθήσω να ε, συντομεύσω λίγο τις απαντήσεις, γιατί και οι άλλες ερωτήσεις ήταν ενδιαφέρουσες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερδύναμη, αλλά παρόλα αυτά ακόμα ανίσχυρη. Νομίζω ότι από απάντησα όταν μίλησα για το Αφγανιστάν, ελπίζω ότι ήσασταν παρούσα ή παρόν. Άρα δεν χρειάζεται να απαντήσω πλέον. Τέσσερις ερωτήσεις μένουν ακόμη. Αν στοχεύουμε στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού, απάντησα ήδη, ελπίζω να σας ικανοποίησα. καταλαβαίνετε ότι δεν θεωρώ ότι είναι και ευφυές να κάνει κανείς κάτι τέτοιο. Μη σας ανησυχεί λοιπόν. Δεν θα ήταν καλή ιδέα. Και μπορώ να εξηγήσω σε οποιονδήποτε αν θέλετε ότι το σωστό είναι να στοχεύσουμε στη δημιουργία επαρκών ικανοτήτων μέσα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει κάθε χώρα μέλος αν θέλει να συμβάλλει. τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για το EUTM. Βλέπω το πρόσωπο που έθεσε την ερώτηση δεν είναι πλέον παρόν. Το είπα, αλλά δεν ανεφέρθηκα στη σχέση μεταξύ EUTM και EUNAFOR. Δεν υπάρχει, δεν είναι η ίδια ιεραρχία, αλλά συμφωνεί ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο εάν επιτύχουμε να φτιάξουμε μια Σομαλία που να μην είναι πλέον αποτυχία ως κράτος. Η εξειδίκευση τώρα του ΝΑΤΟ ως στρατηγικού εταίρου εγώ υποστηρίζω βέβαια την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Άμυνας που λέει βασικά δύο πράγματα. Αφενός αναγνωρίζει και μάλιστα είναι και μέσα στα καθήκοντά μου, στι αρμοδιότητέ μου. Αναγνωρίζει λοιπόν ότι για τι περισσότερε χώρε μέλη το ΝΑΤΟ παίζει σημαντικό ρόλο για την ε, αμυνά του, την ασφάλειά του, αναφέρεται στον διατλαντικό σύνδεσμο κλπ. Ταυτόχρονα προβλέπω, και το είχαμε στο παρελθόν και θα το έχουμε και στο μέλλον, καμιά φορά λοιπόν και κρίσεις Γιατί δεν είναι λογικό το ΝΑΤΟ να έρχεται να λύνει το δικό μα πρόβλημα, διότι είτε πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόβλημα, είτε πρόκειται για ευρωπαϊκό συμφέρον. Δεν μπορούμε να δεχθούμε, ή μάλλον να μην υποδεχθούμε, δεν μπορούμε καλύτερα να αναμένουμε πάντοτε ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα κατανοήσουν για ποιο λόγο πρέπει να έρθουν να λύσουν ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, εφόσον η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει αρκετά για να το λύσει. Θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει μια εύλογη ισορροπία. Και νομίζω ότι ακόμα η ισορροπία δεν είναι κατάλληλη, δεν είναι σωστή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σπαταλά χρήματα μέσω των αμυντικών προπολογισμών, διότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Έχουμε πολλά, ε, ε, πολλούς τομείς ακόμα που ε, μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο. Και επειδή τώρα μειώνονται αναγκαστικά οι προπολογισμοί, και εμένα δεν μου αρέσει βέβαια αυτό, ε, Όμω, ξεπηδάει η ανάγκη να γίνει στενότερο συντονισμός και άρα να δαπανώνται τα όσα χρήματα έχουμε καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Δεν νομίζω θα προχωρούσα σε μια εξειδίκευση μεταξύ ΝΑΤΟ, το ότι το ΝΑΤΟ δηλαδή αναλαμβάνει το στρατιωτικό σκέλος και η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση το πολιτικό. Σύμφωνα και με τη στρατηγική μα, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε την ικανότητα να επιλύσουμε περιφερειακά προβλήματα κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνοι μας ή τουλάχιστον να μπορούμε να πράξουμε τόσα ώστε να είναι πλέον αποδεκτό και από πλευρά άλλων μη ευρωπαϊκών ή μη ενωσιακών χωρών να έρθουν να μας βοηθήσουν διότι θα αντιληφθούν ότι ε, δαπανούν τότε με αποτελεσματικό τρόπο τα χρήματά τους. Αν ε, ε, πιο πιο σημαντικό σε σχέση με την συνολική προσέγγιση, αυτός είναι ο στόχος μας. Παράδειγμα, Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Ηνωμένε Πολιτείε. Μας βλέπουν ως σημαντικό εταίρο. Γιατί? Διότι μιλούν μαζί μου, εφόσον πρόκειται για στρατιωτικό θέμα, γιατί ε, γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτό το μέγα, μεγάλο μέρος ε, ε, ε, σύμπραξης με τον μη στρατιωτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην σχολιάσω καλύτερα για τις πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ αφού ξεφεύγουν απολύτως από τις αρμοδιότητές μου. Αλλά απλώς παρακολουθώ τα τεκτενόμενα ως ε, ε, εμπειρογνώμων που ενδιαφέρεται ειδικά για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα θέματα ήταν πολλά. Θα ρίξουμε ιδιαίτερο φως στην αποστολή κατά της πειρατείας αλλά και για την Σομαλία συνολικότερα καθώς επίσης σχέση μας με τον ΝΑΤΟ και η ε, συνεργασία μεταξύ στρατηγικού και πολιτικού τομέα κυρίως στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης ελπίζω να συμφωνήσετε να σας προσκαλούμε ε, ανατακτά διαστήματα να έρχεστε να μας ε, ενημερώνετε. Σας ευχαριστώ στρατηγέ μου. Bien, nous allons euh, poursuivre avec le deuxième point de notre... Euh, Ερχόμαστε στο θέμα υπαριθμών 2 της ημερήσιας διαταξής μας και με χαρά μας δεχόμαστε, υποδεχόμαστε μάλλον τον ε, Πιέρ Σιμόνοβιτς, υφυπουργός του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας. Η Κροατία η οποία όπως γνωρίζετε ε, είναι αντεπόρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η υποψήφια χώρα η οποία έχει προχωρήσει περισσότερο στον δρόμο της ένταξης. Η Κροατία έχει βέβαια και μακρά ιστορία ε, συνεργασίας ε, και στην άμυνα και ασφάλεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η Κροατία έχει συμμετάσχει κατ' επανάληψη σε επιχειρήσεις και στρατιωτικές και πολιτικές και στην EUFOR στο Τσάντ. Επίσης η Κροατία συμμετέχει στην ΕΟΠΟΛ στο Αφγανιστάν, στο Κόσοβο, στην Αταλάντη και στην Αλθέα, στη Βοσνία, όπου έχει ε, αναλάβει την επιμελητία. Επίσης συμμετέχετε σε άλλες επιχειρήσεις με ελικόπτερα στην μάχημη ομάδα με Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία και την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Από την άποψη λοιπόν αυτή η Κροατία η οποία μας εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2009 γνωρίζει την ε, ε, κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Ε, άλλωστε εσεί επισκεφθήκατε πρόσφατα τον Σέρβο Υπουργό Άμυνα. Είναι σημαντικό οι χώρες οι οποίε επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοικειωθούν με τις ε, δομές ασφάλειας της Ένωσης. Επίσης ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε χώρες οι οποίες υπήρξαν ας πούμε καταναλώτριες των ευρωπαϊκών προσπαθειών ασφάλειας γίνονται τώρα παραγωγή ασφάλειας. Ε, σαφή σταθεροποιητικό ρόλο. Θα εγγύψουμε στα θέματα αυτά. Εξάλλου, σε σχέση με τις σχέσεις σας με τις υπόλοιπες χώρες της ε, περιοχής σας, μίλησα για την επίσκεψη σας στον ε, Σέρβο Υπουργό, επίσης με τη Δημοκρατία της Σερβίας έχετε υπογράψει συμφωνία που καλύπτει ε, θέματα συμφιλίωσης ε, και βεβαίως με τα βλέμματα σταμένα στο μέλλον και έχει ρόλο υποδειγματικό η συμφωνία αυτή ε, με την Σερβία. Έχετε το λόγο κύριε Υφυπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πραγματικά είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο για μένα το ότι μπορώ να συμμετέχω στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πραγματικά προσωπική χαρά. Είναι προνόμιο επίσης, όπως είπα. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με εκφράζοντας θερμότατες μου ευχαριστίες ε, σε εσά και στη χώρα που εκπροσωπείτε, η οποία μας ε, στήριξε για πολλά χρόνια ε, στήριξε την πρόταση για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως ξέρετε είμαστε πλέον στο τελικό στάδιο το προενταξιακό. Έχω ανοίξει 33 κεφάλαια, 22 εκ των οποίων άνοιξαν και έκλεισαν προσωρινά. Άρα πραγματικά είμαστε στη διαδικασία να γίνουμε το σταμότερο δυνατό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε επίσης ότι και εμείς από τη δική μας πλευρά, όπως πράταμε και πράττουμε έτσι και στο τέο μέλλον θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάθε ε, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλους όσους μας έχουν υποστηρίξει. Σε ό,τι αφορά την πολιτική άμυνας και ασφάλειας, την ΚΕΠΑ, που αποτελεί αναπόσπεστο τμήμα και μάλιστα είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι της ε, εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ε, άμυνας. Σε πολλούς ε, τομείς έχουμε ήδη ε, ενσωματώσει την πολιτική σαν να είμαστε ήδη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος ανέφερε τις τάσεις, τις σημαντικότερες τάσεις Συγκεκριμένα πρόκειται για τη συμμετοχή μας σε ειρηνευτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά εκεί η συμμετοχή μας κάνει όλη τη διαφορά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ακριβώς από αυτό το σημείο θα ήθελα να ξεκινήσω. Θα ήθελα να κάνω μια επισκόπηση του πώς αναπτύσσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ε, ΚΕΠΑ. Και όλα θα έλεγα ότι ξεκινούν με αυτό που ουσιαστικά έχει τη μεγαλύτερη σημασία, τον τομέα των επιχειρήσεων δηλαδή. Ήδη από την αρχή συμμετείχαμε στην επιχείρηση U4 για το Τσάντ με 15 μέλη ειδικών δυνάμεων που είχαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν την πολύπλοκη μετάβαση Τη επιχείρηση από την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αιγίδα του ΟΗΕ. Πρόσφατα, με ναυτικούς αξιωματούχου έχουμε συμμετάσχει και σε επιχειρήσεις ε, της ε, επιχείρησης της ακτής Σομαλίας, ε, Γάλλοι, Βέλγοι, Ιταλοί, Ολλανδοί, είχαν στείλει σκάφη και συνεργαστήκαμε και με Ισπανούς συναδέλφους. Και επίσης παρήχε υποστήριξη και ο ναυτικός εξωματούχος μας ε, από το αρχηγείο του Νόρφολκ. Επίσης ε, διαθέτουμε αστυνομικούς ε, για τη Γιούπολ την αποστολή στο Αφγανιστάν καθώς επίσης και μέλη του Υπουργείου Δικαιοσύνης συμμετέχουν στην επιχείρηση Ιουλέξ. Και δωρεάν επίσης ε, είχαμε συμμετάσχει με δύο APC στη Ιούλεξ στο Κωσυφοπαίδιο. Τώρα, ποια είναι η μακροχρόνια δέσμευσή μας. Θέλουμε να παράσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για την ενίσχυση των μόνιμων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέλουμε να συμβάλλουμε στις ομάδες μάχης, τα battle groups της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δεύτερο ήμιση του 2011 θα συμμετέχουμε με 250 στρατιώτες ε, στην ομάδα της επεσηγείται η Γερμανία, ενώ επίσης αποφασίσαμε να συνεισφέρουμε με δύο ελικόπτερα και 20 στρατιώτες για την βόρεια Bell Group που θα είναι επιχειρησιακή στο πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτους, όπως μας ζητήθηκε από τους ίδιους εταίρους που είχαν κάποιες, ε, κάποιες ε, κρίσιμες ελλείψεις στο τομέα των ελικοπτέρων. Και συμφωνήσαμε να τους παρέχουμε τα δέοντα. Όλα αυτά σας τα λέω για να καταλάβετε πόσο βαθιά είναι η συμμετοχή μας ε, στις προσπάθειες αυτές. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ και από τη θέση αυτή αναπτύσσουμε τις δυνάμεις μας ως μια ενιαία δέσμη, ως μια ενιαία δύναμη που μπορεί να υπηρετεί και τις δύο οργανώσεις. Και αυτό που βέβαια έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να μπορούμε να συμμετέχουμε στις επιχειρήσεις σε σχέση με τις ε, συμμετοχές μας στα Battle Group και σε επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαμε σε όλες τις συναντήσεις με την ε, Τρόικα, με την Κομισιόν, ε, όπως και τα άλλα υποψήφια κράτη. Γνωρίζετε την απόφαση της Λέδη Άστον ότι οι, οργανώσεις, οι αυτές οργανώνονται όχι στο περιθώριο όπως γινόταν μέχρι τώρα των οργανώσεων των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, αλλά να είναι ξεχωριστές οι συναντήσεις αυτές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης αναπτύσσουμε τα μέσα για τη συμμετοχή μας ε, στις συνέργειες Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, συμμετέχοντας ε, στην ομάδα δυνατοτήτων ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει ότι μας ενδιαφέρει και το νέο στρατηγικό δόγμα και θέλουμε να είναι πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην ανάγκη σφυριλάτησης ε, πολύ στενή συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο οι δύο αυτοί οργανισμοί να μπορούν να συνεργάζονται από κοινού και στενά μεταξύ τους ώστε να αποφεύγονται αχρίαστες και επιβλαβείς επικαλύψεις και διασπαθήσεις πόρων. Και νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν διάφορα σενάρια στα οποία χρειάζεται ανάπτυξη δυνάμεων. Ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζουμε όλοι σημαντικούς περιορισμούς στους αμυντικούς μας προπολογισμούς. Έτσι λοιπόν, δύο οργανισμοί οι οποίοι μοιράζονται κοινέ αξίες και κοινά μέσα πρέπει να έχουν όλο και πιο στενή συνεργασία μεταξύ τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, την ανάπτυξη των πολιτικών εδώ στις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά άλλες πτυχές της ένταξής μας στην ΚΕΠΑ, ένα σημαντικό στοιχείο του τι συμβαίνει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας είναι ότι η αμυντική μας βιομηχανία, εθνική αμυντική βιομηχανία της Κροατίας είναι καλά ενταγμένη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, που πρέπει να αποτελέσει ένα ουσιώδη στοιχείο για ένα συνολικό αμυντικό μηχανικό πεδίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ό,τι αφορά τον αμυντικό μας σχεδιασμό, και θα έλεγα ότι ουσιαστικά αντικατοπτρίζει αυτός τον αμυντικό σχεδιασμό πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε λοιπόν σημαντική αύξηση της ανάγκης ε, κοινής χρήσης ε, των πόρων, θέσπισης ε, συμφωνιών επιμερισμού του κόστους, επιμερισμού των βαρών, ένας πιο πολυκρατικός χαρακτήρας δηλαδή στον τομέα των αμυντικών βιομηχανιών, των όπλων δυνάμεων, της ανάπτυξης ορισμένων συγκεκριμένων δυνατοτήτων που εξακολουθούν να είναι αναγκαίες για την ε, εθνική και διεθνή ασφάλεια. Συγχρόνως όμως, όταν δεν μπορούν ε, κάποιες από αυτές να τις αναπτύξουν ορισμένες χώρες από μόνες τους, βλέπουμε ότι είναι από πολιτικής πλευράς αναγκαίο χώρες οι οποίες έχουν τις ίδιες αξίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ίδιες απειλές αστάθεια, η διάδοση όπλων, βιολογικός, ακνολογικό πόλεμος, ε, τρομοκρατία. Πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, διότι δεν πρόκειται για απειλές που ε, απευθύνονται μόνο σε μια συγκεκριμένη χώρα, αλλά είναι γενικές απειλές και οι πιο σημαντική απάντηση σε ένα τέτοιο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Έχει να κάνει αυτό και με την οικονομική κρίση. Είδαμε ότι αυτό είχε ω αποτέλεσμα περιορισμού και περιορισμού και αμυντικούς αμυντικού προπολογισμού. Όλα αυτά λοιπόν θέλω να πω ότι μα οδηγούν προ την κατεύθυνση τη συνένωση πόρων, τη συνεργασία του επιμερισμού των βαρών και τις σχετικές ρυθμίσεις. Σε ό,τι αφορά ορισμένες πτυχές της πολιτικής συνεργασίας στην περιοχή, ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, ε, ίσως θα σας ενδιέφερε να ακούσετε ποια είναι η αξιολόγησή μας για το πώς πηγαίνει, ε, πώς θα πηγαίνει η περιοχή και για το ποιες είναι οι πολιτικές μας προτεραιότητες στην περιοχή. Και σε ό,τι αφορά το πρίσμα του Κρατικού Υπουργείου Άμυνας. Πρέπει να σας πω ότι η περιφερειακή και πολυκρατική πολυεθνική ε, συνεργασία είναι ε, ουσιώδης πτυχή της πολιτικής μας και μεταφράζεται σε μία δέσμη αμυντικών συμφωνιών που έχουμε συνάψει με γειτονικέ χώρες. Αναφέρατε εσείς την τελευταία της αμυντική συνεργασία με την ε, Δημοκρατία της Σερβίας κάτι που αποφάσισε το Υπουργείο Άμυνα τη χώρας μου. Έχουμε επίση και άλλε συνεργασίε με πολυμερείς ε, οργανισμού με το χάρτη. και πρέπει να σας πω ότι αυτά τα οποία επιτυγχάνονται στην ευρύτερη περιοχή είναι αποτέλεσμα του των συντονισμένων προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, του ΝΑΤΟ, αλλά και των αμονωμένων χωρών της περιοχής, οι οποίες έχουν ξεπεράσει το παρελθόν, έχουν κλείσει ορισμένα κεφάλαια και έχουν προχωρήσει προς τα εμπρός. Και υπό αυτήν την έννοια υπάρχει και στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών αμυντικών φορέων. Και αυτό σίγουρα ενισχύει και την ευρωπαϊκή σταθερότητα. Ο κινητήριος μοχλός, ή ένας από τους κινητήρους μοχλούς, που ουσιαστικά φέρνει κοντά τις ε, χώρες ε, αυτές είναι το κοινό όραμα του να αποτελούν όλες μια ευρωπαϊκή οικογένεια εθνών. Στις χώρες όλες αυτές οι οποίες θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που με το δικό της ρυθμό η καθεμία προσπαθεί να εκπληρώσει τα απαραίτητα πρότυπα, να προβεί στις ε, απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να προσχωρήσει με την αξία της και με βάση τις φιλοδοξίες της καθεμίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε και φυσικά με τα χαρά θα απαντήσω τυχόν ερωτήσεις. Και βέβαια για μια ακόμη φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας αλλά και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε κύριε Πρόεδρε. Ήταν, μια, ήταν ένα μεγάλο προνόμιο. Ο Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιμούνοβιτς. Έχουμε ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι, αλλά θα ήθελα εγώ να σας θέσω ένα γενικό ερώτημα σε ό,τι αφορά ε, στην ε, αντίληψη που υπάρχει στην ίδια την Κροατία για την ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Καταρχάς, είναι κάτι γνωστό, οι Κροάτες δηλαδή έχουν επίγνωση πολιτική αυτή, ότι υπάρχει αυτή η πολιτική, ότι μπορεί να υπάρξουν προστιθέμενε αξίε, ότι η Κροατία ήδη συμμετέχει ουσιαστικά στι δικέ μα χώρε μέλη. Δεν είναι απαραίτητα κάτι το προφανέ. Φαντάζομαι λιγότερο προφανέ θα είναι στην Κροατία. Ή ε, παραδόξω πώ κάποιε χώρε, ε, λόγω και του ιστορικού πλαισίου, του ιστορικού παρελθόντο, να είναι λίγο πιο ευαίσθητε. Και επίση, ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, ποια είναι η από τη κοινή γνώμη, μια νέα χώρα εντό εισαγωγικών είναι, ε, έχει κάποια απήχηση το ΝΑΤΟ ίσως, είναι πιο δημοφιλές, ε, ε, υπάρχει μια πολιτική αντίληψη όμως στα θέματα, μια ευρωπαϊκή αντίληψη στα θέματα ασφάλειας και άμυνας ε, στην Κροατία. Αυτές είναι πολύ γενικές ερωτήσεις. Ο κύριος Φάγγελ ε, επίσης θέλει να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω κλειμένα μας από την Κροατία. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλώς όρισα λοιπόν τον προσκαλεσμένο μας και του ευχήθηκα σύντομα να μπορεί να μας μιλιάει ως ε, εκπρόσωπος πλήρους μέλους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μεγάλο επίτευγμα για την Κροατία το ότι τόσο γρήγορα είσαστε σε θέση να συμβάλλετε στις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται σε διάφορες αποστολές για την διατήρηση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Είδα τα έγγραφά σας, είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακός, εντυπωσιακό το βιογραφικό σας. Και υποστηρίζουμε λοιπόν την συμμετοχή σας, την ένταξή σας, όχι μόνο στο ΝΑΤΟ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θετικό, πιστεύω, που διαρκώς μιλάτε για τη συνεργασία αυτή που μπορεί να σημαίνει η ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλεια των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη. Μία ερώτηση να σας κάνω. Σε ό,τι αφορά το νέο στρατό επαγγελματιών που έχετε πλέον. Είναι οι άνθρωποι. Ενδιαφέρονται, θέλουν να καταταχθούν στι ένοπλε δυνάμει. να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής ενός στρατιώτη. Εμείς στη Σλοβενία έχουμε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τους νέους που κατατάσσονται. Δεύτερη ερώτηση. Πώς αντιμετωπίζετε τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος ενθουσιασμός για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τμήμα της ερώτησης μπορώ και εγώ να το απαντήσω. Οι δημοσκοπήσεις φυσικά δεν ε, λένε τίποτα για τα πραγματικά συμφέροντα, γιατί θεωρώ ότι όταν πρόκειται για πραγματικές αποφάσεις, ο κόσμος λαμβάνει υπόψη τι θα κερδίσει, τι θα χάσει και είναι προφανές ότι οι Κροάτες ξέρουν τα πλεονεκτήματα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά όμως θα ήθελα να σας θέσω την ερώτηση αυτή. Χαίρομαι επίσης, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, βλέποντας την προσέγγιση μεταξύ Κροατίας και Σερβίας, πρέπει να πω ότι ήταν μια πολύ σημαντική διαδικασία η οποία πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο ικανοποιητικό για όλες τις πλευρές και αυτό είναι ιδιαίτερα καλό, ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Ότι ξεκίνησε συνεργασία επίσης και στον στρατιωτικό τομέα. Είναι καλό σημάδι. Και το γεγονός ότι τα πιο πολλά από τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ της Κροατίας και των άλλων γειτονικών χωρών έχουν πλέον είτε ολοκληρωθεί είτε σχεδόν ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα εισαγωγικά σας σχόλια και σας καλωσορίζω ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, κυρία Λονατσέκ. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος και της δικής μου πολιτικής ομάδας θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία μας το συντομότερο δυνατόν να ενταχθεί η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε που ήλθατε και που μας μιλήσατε ως Υφυπουργό για το ποια είναι η θεώρησή σας για την ε, πρόοδο της Κροατίας. Να υποστηρίξω τον Πρόεδρο στην ερώτηση που έθεσε. Η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας πώς γίνεται αντιληπτή στην Κροατία. Δεύτερο ερώτημα σε ό,τι αφορά την ένταξη της Κροατίας στην Ένωση. Διάβασα σήμερα χθε σε κάποια εφημερίδα ότι δυστυχώς η υποστήριξη, μάλλον σύμφωνα με μια δημοσκόπηση, η υποστήριξη λοιπόν του κόσμου για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιοριστεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό. Ξέρω ότι είστε Υπουργό άμυνα, αλλά παρόλα αυτά σα ανησυχεί αυτό. Εμά μα ανησυχεί. Γιατί αν γίνει δημοψήφισμα, δεν θα ήθελα μετά από όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έχουμε περάσει και που έχετε περάσει και εσείς και έχουμε υποστηρίξει να είναι αρνητική απάντηση. Αυτό που μας είπατε επίσης για το ρόλο της Κροατίας και σε θέματα άμυνας. Πριν ε, έλθετε, συνομιλήσαμε με τον αντιστράτηγο Φανός από την Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Επιτελείο και μιλήσαμε για τη συνεργασία πολιτικού και μη πολιτικού σκέλους, ε, στρατιωτικού και μη στρατιωτικού σκέλους. Πώς θεωρείτε ότι αυτό το πολιτικό σκέλος μπορεί να διαμορφωθεί από πλευρά Κροατία. Μιλήσατε για το διευθυντικό σκέλο και είναι αναπόφευκτο αυτό, μια και είστε υφυπουργό άμυνα. Αλλά ξέρετε, γίνεται μια ε, έντονη προσπάθεια σε ό,τι αφορά το μη στρατιωτικό σκέλο, την ε, πρόληψη κρίσεων και το καθεξής. Για τις ομάδες μάχης τώρα, κάποιοι θέλουν να χρησιμοποιούνται και σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό. Θα ήθελα να υπάρξει, για παράδειγμα, μια ομάδα άμεση αντίδραση σε ό,τι αφορά τέτοια θέματα ανθρωπιστική κρίση. Ποια είναι όμω η θέση και τη δική σα κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ο Υφυπουργό έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσει που μου θέσατε. Να ξεκινήσω με αυτά που είπατε εσεί, κύριε Πρόεδρε. Για το πώς γίνεται αντιληπτή η ΚΕΠΑ στην Κροατία και στην ευρύτερη περιφέρεια. Να, να πω ότι χάρη στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της ΚΕΠΑ και της ΕΠΑ, στην περιφέρεια, στην περιοχή μας, για παράδειγμα στη Βοσνία, με την επιχείρηση Αλθέα, η πτυχή της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον ευρέως ε, γνωστή και την εκτιμάει ο κόσμος. αν και βασικός πυλώνας της ασφάλειας παραμένει το ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά την αντίληψη του περισσότερου κόσμου για την άμυνα, για το στρατιωτικό σκέλος. Εκ παραλλήλου όμως, υπάρχει και επίγνωση του τι σημαίνει η συνθήκη της Λισαβόνα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη ρήτρα αλληλεγγύης και το τι συνεπάγεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το στρατιωτικό της σκέλος ε, η συνθήκη της Λισαβόνας. Και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες σε επίπεδο κυβερνητικό. Γίνονται πολλά σεμινάρια, διασκέψεις για τους ε, αξιωματούχους διάφορων υπουργείων προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα για την ΚΕΠΑ, να ενημερωθούν για τις πολιτικές Άρα είναι όλο και πιο αυξανόμενοι, αν θέλετε, όλο και πιο πολλέ γνώσει υπάρχουν για το θέμα αυτό. Και στην Κροατία και στην ευρύτερη περιοχή. Και η συμβολή όλων των χωρών στις διάφορες επιχειρήσεις έχουν γίνει πολύ γνωστές και αυτό δεν ισχύει μόνο για την ε, Κροατία αλλά και για τους Σέρβους ομολόγους μας. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τσάντ. Άρα, είναι ευρέως γνωστό το τι κάνει κάθε χώρα σε κάθε επιχείρηση. και όλο και πιο πολλοί κόσμος γνωρίζει και την ευρωπαϊκή διάσταση, τη διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις αυτές. Σε ό,τι αφορά, κυρία Λούνα, τσεκ την ανάπτυξη του μη στρατιωτικού σκέλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει καταλάβει την αρμόζουσα θέση στην όλη αντίληψή μας. Έχουμε και δικαστικούς, διπλωμάτες και την γενικότερη αντίληψη ότι υπάρχει η ανάγκη αυτή, η επιτακτική του μη στρατηγικού σκέλους για πολλά καθήκοντα τα οποία πρέπει να αναλάβει το πολιτικό σκέλος αυτό. Και υπάρχει ένας ευρύτατος τομέας για την ε, ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μάχημες ομάδες. Ξέρετε ότι συμμετέχουμε σε δύο εξ αυτών. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει ένα ε, εργαλείο λειτουργικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η έννοια της μάχημης ομάδας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για την λειτουργικότητα του μέσου αυτού. Για διάφορα σενάρια. Συμφωνώ ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται αυτές οι ομάδες για οποιοδήποτε σκοπό. Υπάρχει και ένα οικονομικό, ένα και ένα οικονομικό σκέλος. Σε ό,τι αφορά όμως ε, την αστάθεια του διεθνού ε, προσκηνίου θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι ομάδες. Κύριε Βάγκελ, σε ό,τι αφορά το πόσο ελκυστικό είναι το επάγγελμα του στρατιωτικού στην Κροατία. Δυστυχώ, μάλλον ευτυχώ, ε, προσελκύουμε το ενδιαφέρον των νέων. Κατατάσσονται πολλοί κόσμος. Και αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει αντίληψη ότι έχουν αλλάξει οι ένοπλες δυνάμεις, ε, ότι είναι πιο σύγχρονες, έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, προσεγγίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρόκειται για ένα ενδιαφέρον ε, επάγγελμα, μία ενδιαφέρουσα καριέρα. Το οποίο συνεπάγεται εξειδίκευση, εκπαίδευση, κατάρτιση, ε, αξιώματα στο εξωτερικό, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά υπάρχει και ο οικονομικός παράγοντας. Και γι' αυτό λοιπόν είναι όλο και πιο δημοφιλές ε, το επάγγελμα. Προσελκύουμε πολλούς νέους λοιπόν. Χάρη και στο σύστημα εθελοντικής κατάταξης. Δεχόμαστε δηλαδή ομάδες ε, ατόμων, οι οποίοι μπορεί να μην είναι τελικά επαγγελματίε στρατιωτικοί. Μπορεί μετά από κάποια εκπαίδευση να αποφασίσουν ότι θέλουν να μείνουν, μπορεί και όχι. Προσελκύουμε λοιπόν επαρκές ενδιαφέρον. Προσελκύουμε αρκετούς νέους. σε ό,τι αφορά την αντίληψη που επικρατεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ο διάλογος με το κοινό για όλες τις ευθύνες και όλα τα πλέον εκτήματα που σας συνεπάγεται η ένταξή μας στην Ένωση είναι σημαντικός. Αυτός όμως ε, γίνεται ο διάλογος και γίνεται σε όλη τη χώρα και σε όλα τα επίπεδα του πληθυσμού, σε όλα τα επίπεδα του κόσμου, γιατί όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποιος θα είναι ο αντίκτυπος θα πρέπει λοιπόν με σωστό τρόπο να τους εξηγήσουμε το θετικό χαρακτήρα των συνεπειών. Διαρκώς λαμβάνουμε αποτελέσματα δημοσκοπήσεων όπου αναφέρεται ότι ο κόσμος κατά 60% τάσσεται υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που και που υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων με διαφορετικά αριθμητικά αποτελέσματα αλλά όλα, α, ξέρετε, εξαρτώνται από τον τρόπο που τίθεται το ερώτημα ή αν θέλετε από την ημέρα που έχει διεξαχθεί το η δημοσκόπηση. Η τάση είναι θετική πάντως. Όταν θα γίνει γνωστή και η ημερομηνία για την υπογραφή των πρωτοκόλων ένταξης, όταν θα γνωρίζουμε την ημερομηνία και θα γίνει ίσως ε, δημοψήφισμα, θα διεξαχθεί και ο τελευταίος γύρος του διαλόγου με τον κόσμο. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα σημαντικό τομέα στον οποίο θα μας ε, βοηθούσαν και οι εμπειρίες των δικών σας χωρών. Και τι καλύτερο υπάρχει από το να ακούμε από μια χώρα η οποία πρόσφατα πέρασε την όλη εμπειρία της ένταξης να βγαίνει εκπρόσωπο της χώρας αυτής, να μιλήσεις στο κοινό στην Κροατία και να αναφέρει το τι άλλαξε στη χώρα του. Από τη γεωργία μέχρι τα ναυπηγεία. Για όλους τους τομείς του πληθυσμού. Συνολικά όμως πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι η τάση είναι θετική και είμαστε αισιόδοξοι ότι όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα είναι σαφής η απάντηση και θετική. Ευχαριστώ πολύ. Αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να σα κάνω δύο ερωτήσει που ίσω να μην έχουν άμεση σχέση με αυτά που αναφέραμε μόλι πριν. Αφορούν όμω και τη χώρα σα και την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Το πρώτο είναι το εξή. Μιλήσαμε για τη γαλλο ρετανική Συμφωνία σε θέματα άμυνα στην προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Θεωρείτε εσεί ότι είναι ίσω μια αγωιστική προσπάθεια των δύο χωρών που έχουν ανώτερε δυνατότητε και που τελικά ξεκινούν μόνε του ε, ε, μια συγκεκριμένη πορεία, ή μήπω θεωρείτε ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να ε, φέρει κοντά και άλλε χώρε που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα, θα είναι ένα είδο ηλεκτροσόκ δηλαδή για τι άλλε χώρε. Το δεύτερο ερώτημα. Ξέρετε ότι εμεί στο Κοινοβούλιο παρακολουθούμε κάποια που μας πολύ στενά τη διαδικασία προσχώρηση τη Κροατία. Είχε έρθει και ο εισαγγελέα ε, Μπραμέρτ εδώ πριν από κάποιου μήνε, ο οποίο είχε εκφράσει κάποια παράπονα. Τέλο πάντων, είχε πει ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν ε, με την Κροατία σε ό,τι αφορά την τεκμηρίωση, τα έγγραφα. Ποια συνεργασία, τι συνεργασία ε, υπάρχει, δηλαδή το Υπουργείο Άμυνα, τη Κροατία, πώ συνεργάζεται με τη Χάγη και τι μπορείτε να μα πείτε για αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσει, κύριε Πρόεδρε. Για το πρώτο θέμα, για την αμυντική συνεργασία, στο παράδειγμα αυτής της ε, Entente Κορδιάλ, αν μπορώ να την πω έτσι, μεταξύ των Γάλλων και Βρετανών φίλων μας, αυτό ασφαλώς είναι κάτι το οποίο ε, αξίζει να υποστηριχθεί και είναι σωστός δρόμος. Σε ορισμένους τομείς όπου υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όπου δεν θέτει σε κίνδυνο την συνολικότερη αρχιτεκτονική της Ένωσης. Εμείς βέβαια δεν είμαστε ακόμη μέλη, αλλά παρακολουθούμε εκ των έξω. Έχει ενδιαφέρον να υπάρχουν ορισμένες ομάδες που να προηγηθούν σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία ε, και την εξέβρεση πολυεθνικών λύσεων. Θεωρούμε ότι αυτό είναι αναγκαιότητα. Εμείς ήδη θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τέτοιους μηχανισμούς. Υπάρχει ένα φάσμα αμυντικών ικανοτήτων, αμυντικών ε, δυνατοτήτων που πρέπει να διαθέτουν οι χώρες μέλη. Ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς των αμυντικών προϋπολογισμών, καμιά χώρα δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη της. Άρα η λογική συνέπεια της σκέψης αυτής είναι να υπάρξει μια ε, κοινή προσπάθεια, ένα pooling and sharing, όπως λένε στα αγγλικά. Για άλλες χώρες ίσως να μην είναι βέβαια τόσο εύκολο εφαρμοστεί αυτό. Υπάρχει πάντως γνήσιο ενδιαφέρον από πλευράς πολλών χωρών και εμείς θεωρούμε ότι αξίζει να ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος χωρίς όπως είπα να τεθεί σε κίνδυνο η ενότητα ε, του συνόλου. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στον ίδιο δρόμο στη συνεργασία με τους εταίρους μας. Εξάλλου, Έχουμε κάνει και με συνέπεια όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να ικανοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις του δικαστηρίου της Χάγης και του κ. Μπράμερτς με ομάδα ειδικών καθηκόντων που έχει δημιουργηθεί και που ε, υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που μας συζητήθηκαν και μάλιστα υπάρχει και μια σειρά από διαδικασίες και δίκες που έχουν προχωρήσει σε βάρος ατόμων με, με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκριθούμε στα όσα απαιτούνται από εμάς και αυτό έχει γίνει δεκτό από τους εταίρους μας και εμείς θα συνεχίσουμε. Ή εν πάση περιπτώσει το Υπήρξαν ορισμένες καταγγελίες σχετικά με ορισμένα έγγραφα, τα οποία ίσως να υπάρχουν, ίσως και να μην υπάρχουν. Και ένα από τα καθήκοντα αυτής της ομάδας, ιδιαίτερων καθηκόντων της Task Force, ήταν και αυτό. Άρα, ορισμένα έγγραφα δεν υπάρχουν Όσα πάντως ε, υπάρχουν έχουν υποβληθεί και δεν έχουμε φυστεί προσπαθειών για να τα ε, διαβιβάσουμε στην Χάγη. Άλλωστε θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή και μέχρι τέλους. Η κυρία Λούνατσεκ, ευχαριστώ και ε, Υπουργέ, δύο ακόμη θέματα ίσως έχει ενδιαφέρον να σας ρωτήσω. η ένταξή στον στο ΝΑΤΟ συνεπάγεται και σημαντικό κόστος για τον προϋπολογισμό σας. Υπήρξαν, τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο μπορέσατε να αντιμετωπίσετε εύκολα, το αντιμετωπίσατε ήδη. Και πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη στην χώρα σας, αφού και εσείς βρίσκεστε μέσα στην κρίση όπως όλοι. Άκουσα και κάποιες ιδέες για μια κοινή αεροπορική άμυνα μεταξύ Ιταλίας, Σλοβενίας και Κροατίας. Ε, περί τίνος πρόκειται. Σας ευχαριστώ κυρία μου για την πρώτη σας ερώτηση. Ασφαλώς και εμείς έχουμε σημαντικούς περιορισμούς ό,τι αφορά μια ενδεχόμενη αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού μας το ιδεώδες θα ήταν να είχαμε φτάσει το 2% του ΑΕΠ μας, αλλά για την ώρα βρισκόμαστε στο 1,37%. Ο προπολογισμό μας λοιπόν πράγματι δεν κατέστη δυνατόν να αυξηθεί σύμφωνα και με τις προηγούμενες οικονομικές προβλέψεις. Ό,τι αφορά τώρα την σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και αμυντικού προπολογισμού, και αυτό νομίζω εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντασσόμαστε σε μια συμμαχία. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε όλες τις αμυντικές ικανότητες όπως θα έπρεπε αν ήμασταν μόνοι μας. Θα ρίξουμε το ιδιαίτερο βάρος λοιπόν στα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και για τα υπόλοιπα αναμένει κανείς από τους συμμάχους να καλύψουν τις ανάγκες. Ενώ βεβαίως και εμείς από τη δικιά μας μελπρεβά κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο και ό,τι αναμένεται από εμάς. Εν τέλει η θέση μας θα είναι καλύτερη όντας ενταγμένοι στο ΝΑΤΟ από ό,τι αν ήμασταν μόνοι μας. Και βεβαίω, τελικά ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας θα είναι πολύ μεγαλύτερος μέσα στην ένταξή μέσω της ένταξή της μάλλον. Βρίσκουμε λοιπόν θετικό το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ από την άποψη αυτή. Και βέβαια βοηθεί αυτό ώστε να, μια χώρα να εξετάσει ποικίλε πολυεθνικές λύσεις οι οποίες τη επιτρέπουν να εξοικονομήσει κάποια πράγματα και να κάνει ορθολογητικότερη χρήση των πόρων της. Επίσης, ο Σλοβαίνος και Κροάτης Πρωθυπουργοί δήλωσαν ότι θα εξετάσουν τρόπους για μια ενδεχόμενη συνεργασία στους εθέρες. Ακριβώς μέσα σε αυτήν την ανάληψη κοινών βαρών και στην ένταξή μας σε πολυεθνικές λύσεις, που είναι μια τάση που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δείχνει και το γαλλοβρετανικό παράδειγμα, που θα μας οδηγήσει η προσπάθεια αυτή, ακόμα δεν το γνωρίζουμε, αλλά πάντως αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να συζητήσουμε και αυτά αλλά και άλλα θέματα με τους Σλοβαίνους φίλους μας, να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να αποφύγουμε επικαλύψεις, πώς μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή την κοινότητα ενδιαφερόντων και συμφερόντων που έχουμε με τους Σλοβαίνους. Προσωπικά έχω έρθει σε επαφή με τους Σλοβαίνους φίλους μας νομίζω θα συζητήσουμε και άλλους τομείς συνεργασίας και βεβαίως η ε, άμυνα στον αέρα είναι ένας από τους τομείς. Τώρα και οι δύο χώρες μας είναι ε, στο ΝΑΤΟ. Είναι ενταγμένες στα συστήματα ραντάρ του ΝΑΤΟ. Για την ώρα υπάρχουν βέβαια ξεχωριστές αρμοδιότητες και ευθύνες αστυνόμευσης των εθέρων κλπ. Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να συντεριάξουμε τα, τις, τις αμυντικές μας ανάγκες με κάποιες εξοικονομήσεις και ταυτόχρονα τα αμυντικά μας ε, συστήματα να συμβάλλουν ώστε να διευκολυνθούν και να προαχθούν ακόμα περισσότερες σχέσεις μεταξύ των χωρών μας. Τα θέματα αυτά αξίζει τον κόπο να συζητηθούν με τους Σλοβαίνους όπου και να οδηγήσουν οι τέλει. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας. Όπως θα διαπιστώσατε όλες οι πολιτικές ομάδες και τις που... Um, uh, well, I think the, main help is probably whilst legislation is still being developed in Europe. I think once it's passed, we're often behind the game. Um,